más tarde, por la mañana Good day. Good day everybody. Good morning. Καλημέρα σας. Work. We had a long day yesterday. Χθες είχαμε πραγματικά μια μακριά και κουραστική μέρα, το ίδιο και σήμερα. Έχουμε και πρωινή και απογευματινή συνεδρίαση και θα ξεκινήσουμε με το σημείο 12 που προβλέπει κοινή συνεδρίαση τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Πολιτικών Ελευθεριών για το πρόγραμμα δικαιοσύνη για την περίοδο 2014-2020. Θα γίνει μια παρουσίαση της σχέδιας έκθεσης σε ό,τι αφορά την πρόταση κανονισμού για το πρόγραμμα δικαιοσύνη περίοδος 2014-2020. Έχουμε δύο συνεισηγητές εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, τον κύριο Φίλιπ Κλέης και εκ μέρου τη επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έχουμε τον κύριο Λουίτζι Μπερλιγκουέρ. Όπως ξέρετε... With the, uh, Προβλέπεται η συνηθισμένη νομοθετική διαδικασία με συνεργασία βάσει του κανόνα 51 δύο επιτροπών της ΛΥΜΠΕ και της ΓΙΟΥΡΙ. Γι' αυτό έχουμε και έκθεση με δύο συνεισηγητές έναν από κάθε επιτροπή. Πριν τους δώσω το λόγο, θα ήθελα να σας πω ότι η προθεσμία για την κατάθεση των ροπολογιών λήγει στις 5 Ιουλίου το μεσημέρι, 12 η ώρα. Η εξέταση των τροπολογιών θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Καστέξ, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Καλώς ήρθατε κυρία Κάστεξ. Θα μας κάνετε μια εισαγωγή και μετά θα μας παρουσιάσουν οι δύο συνεισηγητές τα σχέδια εκθεσής τους. Η κυρία Καστέξ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Λόπες Αγγελάρ, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτά που μας είπε ο πρόεδρος Λόπες Αγγιλάρ. Ο φάκελος αυτός είναι η επιβεβαίωση και η συνέχεια μιας πολύ αγαστής συνεργασίας μεταξύ της Νομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών που κρατάει εδώ και πολύ καιρό. Το πρόγραμμα αυτό είναι ο διάδοχος και η φυσική συνέχεια τριών προηγούμενων προγραμμάτων της πολιτικής δικαιοσύνης, της ποινική δικαιοσύνης και το πρόγραμμα της πρόληψης α, ε, χρήσης ναρκωτικών και της ενημέρωσης του κοινού. Πρόκειται για ένα θεμελιώδες εργαλείο για την προώθηση της δικαστικής συνεργασίας σε θέματα ε, αστικού και ποινικού δικαίου για την περίοδο 2014-2020. Φυσικά θα πρέπει με επαρκή κονδύλια να χρηματοδοτηθούν από την κοινότητα κάποια προγράμματα προκειμένου να εφαρμοστούν οι πολιτικές και νομοθετικές ε, αποφάσεις στον τομέα της δικαιοσύνης ε, με ιδιαίτερη εστίαση στα διασυνοριακά θέματα που, χρήζει, που χρήζουν συντονισμένη συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το δημοσιονομικό κονδύλιο που προβλέπεται από την, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα αυτό είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό δεν μπορεί να τροποποιηθεί από τις τροπολογίες σας. Και στα πλαίσια ε, του πολιτου δημοσιονομικου δημοσιονομικού προγράμματος 2014-2020 αυτά τα 472 εκατομμύρια που προβλέπονται ε, θα ε, δεν εμπίπτουν, επαναλαμβάνω, στις τροπολογίες. Οι δύο, τροπο, δύο επιτροπές θα πρέπει να τροπολογήσουν κάποιες δράσεις ίσως του προγράμματος της δικαιοσύνης για να βελτιωθεί η διαφάνεια, η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα αυτού του προγράμματος. Αυτό το αφήνω στη δική σας ε, οξυδέρκεια και της, την ευρηματικότητα για την υποβολή τροπολογιών. Πάντω η έκθεση αυτή είναι πολύ συγκροτημένη, μεστή, πολύ ικανοποιητική και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους δύο συνεισηγητές, τους κυρίους Κλέη και Μπερλιγκουέρ, για το πολύ αξιόλογο όνειμά τους που θα είναι χρήσιμο για όλους και που βελτιώνει αισθητά την πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ θερμά του συνεισηγητέ και ξαναδίνω το λόγο στον πρόεδρό σα, τον κύριο Λόπη Αγγιλάρ, για τη συνέχιση τη συνεδρία Περιμένουμε να πάσει στιγμή και τον κύριο Μπερλιγκουέρ από την Νομική Επιτροπή. Πάντω, ο, Επιτροπής, τη ο Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών είναι παρόν, ο κύριος Κλέης και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το πρόγραμμα για την δικαιοσύνη που είναι και το αντικείμενο της έκθεσής μας, είναι ουσιαστικά η περίληψη τριών προγραμμάτων. Το πρόγραμμα για την η το θέμα της ενημέρωσης και μία σειρά προγραμματικών προτάσεων εμπεριέχονται σε αυτό το πρόγραμμα, όπως οι μη σαφείς διαδικασίες, το θέμα της ε, ευελιξίας. Κανείς δεν ξέρει σήμερα ποιο είναι, αν θέλετε, το προστιθέμενο κέρδος, προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε σχέση με τα εθνικά συστήματα. Η αξιολόγηση δηλαδή της πραγματικής ε, χρήσης, του πραγματικού αποτελέσματος αυτού του προγράμματος. Ο κύριος Μερλιγκουέρ και εγώ προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα αυτά στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου έχουν μια προστιθέμενη αξία, ότι συνεισφέρουν δηλαδή με ένα πολύ σαφή τρόπο στη βελτίωση του συστήματος δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Αυτό βεβαίως μπορεί να συμπεριλάβει κάποιες ε, τοπικές, ε, περιφερειακές ε, πρωτοβουλίες, σεβόμενη την αρχή της επικουρικότητας. Σχέδια λοιπόν τα οποία είναι μικρότερης κλίμακας μπορούν να συμπεριληφθούν. Όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή και την πιο δίκαιη κατανομή, πιστεύουμε ότι ο γλωσσικός παράγοντας μπορεί εδώ να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο και πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στο γλωσσικό τομέα στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε κάποιους από τους στόχους. Ενισχυμένη συνεργασία, παραδείγματος χάρη, όταν υπάρχουν γλωσσικά προβλήματα. Το βασικό έγγραφο, το οποίο έχει συνταχθεί μόνο στα αγγλικά, είναι ένας έμεσος τρόπος να θεωρήσει κανείς, να φτάσει κανείς στο συμπέρασμα ότι όποιος θέλει να συμμετάσχει μπορεί να το κάνει μόνο στα αγγλικά. Όχι, βεβαίως και όλες οι επίσημες γλώσσες εδώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Απλώς το έγγραφο είναι σήμερα διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά. Πιστεύω ότι αυτό πραγματικά μπορεί να έχει κάποιες επιπτώσεις όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή και αυτό κυρίως σε χώρες όπου τα αγγλικά δεν είναι τόσο διαδεδομένα. Υπάρχει λοιπόν μια βασική αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει πάντα να προσπαθούμε όλες τις γλώσσες να τις αντιμετωπίζουμε σε ίσο με σε ίση βάση και βεβαίως η εκμάθηση άλλων γλωσσών είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τους συνεργάτες που εργάζονται στον τομέα της δικαιοσύνης. Όμως, για να υπάρξει πραγματική διαφάνεια για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα κείμενα αυτά σε όλες τις επίλυμες γλώσσες. Εάν θέλουμε αυτό το πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη να είναι ευρέως αποδεκτό. Επίσης, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να υπάρξει και μία μεσοπρόθεσμη έκθεση το 2017 και η τελική έκθεση το 2021. 2021. Θα διπλασιάσουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Υπάρχει σήμερα ο ιστότοπος αλλά θα πρέπει να τον βελτιώσουμε έτσι ώστε να βρίσκει κανείς και όλα τα ονόματα των ε, σχεδίων, αλλά και κάποιες λεπτομέρειες. Βλέπουμε ότι η Επιτροπή δέχεται όλες αυτές τις προτάσεις και αυτό είναι κάτι το πολύ θετικό. Κάτι άλλο που θα ήθελα να υπογραμμίσω. Μία ολόκληρη σειρά σχεδίων και προγραμμάτων μπορούν να καλυφθούν και σε συνεργασία με τους και όδησης διαπιστώσαμε ότι υπάρχει συμφωνία για την ενσωμάτωση κάποιων σχεδίων στο πρόγραμμα αυτό. Όχι βέβαια όλα. Βεβαίως και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε προγράμματα που αποκλείονται σήμερα. Δεν τα αγνοούμε τελείως, αλλά δυστυχώς σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να περιοριστούμε στην ουσία του κειμένου και όχι σε όλες τις επιμέρους πτυχές και τις ιδεολογικές σκέψεις παραδείγματο χάρη. Το θέμα της κατάρτισης είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν εδώ την εντύπωση ότι παραδείγματο χάρη για την καταπολέμηση της χρήσης και της εμπορίας ναρκωτικών Βεβαίως και η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα κονδύλια λοιπόν που διατίθενται σήμερα για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας θα πρέπει να αυξηθούν. Η δράση αυτή πρέπει να ενισχυθεί και το πρόγραμμα για την καταπολέμηση των ναρκωτικών θα πρέπει σαφώς να συνεχιστεί. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο διαθέτει σήμερα πολύ περιορισμένους πόρους σε σχέση με άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 500 εκατομμύρια ευρώ τα οποία βεβαίως θα πρέπει να δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες πώς κατανέμονται και πώς δαπανώνται για να δούμε αν υπάρχει η προστιθέμενη αξία την οποία αναμένουμε. Και βεβαίως θα ακολουθήσει μια αξιολόγηση έτσι ώστε να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή και τον συνάδελφο, τον κύριο Μπελίνγκουαρ από την Νομική Επιτροπή, γιατί πραγματικά είχαμε μια εξαιρετικά επικοδομητική συνεργασία. Ήδη έχουν υποβληθεί <laughs> προτάσεις για τη βελτίωση αυτού του κειμένου και βεβαίως θα τις εξετάσουμε σε λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος ζητάει το λόγο. Ναι, έχετε το λόγο. Θα προεδρεύσω για 10 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως βλέπετε, αν δεν έχετε αντίληψη, θα συνεχίσω και εγώ στα Ολλανδικά, όπως βλέπετε, στην ίδια γλώσσα που και ο προλαλή σα. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και οφείλω να ομολογήσω πως δουλέψαν πάρα πολύ καλά μαζί οι δυο και νομίζω πω οι δύο επιτροπέ μα συμφωνούν σε πολλά σημεία όταν πρόκειται να δούμε τι πιο σημαντικέ πτυχέ αυτή τη εκθέσεω. Ο αντιπρόεδρο τη Νομική επιτροπή μα είπε πω το θέμα δεν είναι να δούμε ποιο είναι το ποσό το οποίο τίθεται, αλλά είναι να μπορέσουν οι δύο επιτροπές να υποστηρίξουν τις δικές τους αρμοδιότητες γιατί η Επιτροπή Προϋπολογισμού και της Γεωργικής και της Περιφερειακής οι συνάδελφοι αυτοί λοιπόν από αυτές τις τρεις επιτροπές έχουν την τάση να δίδουν πολύ μεγάλη σημασία στα νούμερα, στα ποσά και όταν πρόκειται για τη δικαιοσύνη στα πλαίσια της ε, πρέπει να υποστηρίζουμε εμεί ο καθένας το δικό του χώρο. Υπάρχουν ακόμη πολλά στοιχεία τα οποία δεν έχουν ξεκαθαριστεί στα κονδύλια του προπολογισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει πως θα πρέπει να επιμείνουμε ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα εκείνα τα οποία τους έχουν κατανεμηθεί. Ξέρετε υπάρχουν πολλοί νομικοί, ε, εισαγγελείς, δικαστές, δικηγόροι κλπ. Και τα τελευταία χρόνια πολύ περισσότερο επιμείναμε για αυτά τα σημεία, για αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα όμως βρισκόμαστε σε ένα βέλτιστο σημείο, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε μια κατάρτιση δικαστών και δικηγόρων και πολύ περισσότερο επιμένουμε σε κατάρτιση αυτών των δύο τελευταίων. Ο εισηγητής λοιπόν μας μας παρουσιάζει όλες τις πτυχές της νομικής επιστήμης και νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν τα δικαστήρια στην Ευρώπη να μπορέσουν να εκφράζονται επ' αυτών των θεμάτων. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο είναι πολύ καλή ιδέα να προβλέπονται μαθήματα γλώσση. Ο εισηγητή εκ περισσού μα ζητά και μα ζήτησε καλύτερα κατά πόσον δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε με πολύ, πολύ πιο σαφή τρόπο το αίτημα αυτό για περαιτέρω συνεργασία στο θέμα το γλωσσικό. Μου η εντύπωση ότι εξ υπαρχής συμμετέχουμε. Και βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, τα, τα, συγγνώμη, υπάρχουν προγράμματα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω. Και αυτό κατατίθεται ήδη στην προκαταρκτική, στο προήμιο της εκθέσεως, λέγεται πάρα πολύ σαφώς. Και θα πρέπει να δουν πραγματικά τους στόχους οι οποίοι έχουν επιτευχθεί ήδη και αυτούς που θα τεθούν για το μέλλον. Δύο ακόμη παρατηρήσεις, Πρόεδρε για να πω πως συμφωνώ απολύτως με αυτό που ελέγχθη από τον εισηγητή όταν πρόκειται για το θέμα της καταπολέμησης των ναρκωτικών θα πρέπει να επιβιβλούν πολύ περισσότερο στην πρόληψη παρά στην καταστολή και πιστεύω πως το πρόγραμμα αυτό της πρόληψης θα πρέπει να το συλλάβουμε, θα πρέπει να το διαμορφώσουμε, να το εκπονήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να καταπολεμήσουμε αυτό, το πλήγμα. Και υπάρχει ακόμη το θέμα όλων αυτών των πράξεων κατεξιοδότηση. Και νομίζω πως θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσουμε και να δούμε κατά πόσο ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν μπορεί να επιμείνει από αυτό το σημείο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευκοινοβούλιο να μπορεί να εκφράσει την αποψή του θέματο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα την κυρία Ρισμπέκ να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Και ο κύριο Μπερλίνγκο μόλι φτάνει, νομίζω, και θα του δώσω το λόγο αμέσω μετά. Κύριε Ρισβέκ. Κυρία Πρόεδρε, μου δίνετε το λόγο. Και εγώ θα ήθελα από την πολιτική μου ομάδα να, εισηγεί, να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία που έχει γίνει, καθώς επίσης και για το κείμενο της Κομισιόν το οποίο έχει τροποποιηθεί, που αποτελούν τη βάση αυτής της συνεργασίας. Και όλοι το θέλουμε, όλοι το ευχόμαστε και θα υλοποιηθεί με ένα απλό και λογικό τρόπο και ευανάγνωστο τρόπο. Και χρειάζεται βέβαια αυτή, αυτό το κτέλισμα του, του το χτένιμα αυτό του κειμένου για την καλύτερη παρουσίασή του. Όσον αφορά βεβαίω την κατανάλωση των ναρκωτικών. Πριν πω οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να επιμείνω επί του κειμένου, το οποίο εξετάστηκε και από την ομάδα μας και θα υπάρξουν οι τροπολογίες και να επενθυμίσω ότι δεν υπάρχει έψινα ψηλών εάν δεν υπάρχει αυτή η ιδέα της ενίσχυσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ των πολιτών των χωρών. Γιατί αυτό το οικοδόμημα μιας νομικής κουλτούρας, νομικού πολιτισμού αν θέλετε, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ καλά στην εργασία της, του εισηγητού, έχει μια κεφαλαιότητη σημασία σε σχέση με την ενίσχυση της ΕΕ. Υπενθυμίσατε τους όρους των ορίων του προπολογισμού πόσο μας παίρνει στον προπολογισμό, αλλά το πιο βασικό είναι όσον αφορά τη συνεργασία, τη διασυνοριακή. Εγώ μένω σε, κοντά στα σύνορα και γνωρίζω πως εάν αυτή η συνεργασία και αυτός ο χώρος ο δικαστικός, νομικός, πάρει σάρκα και οστά, νομίζω πως πραγματικά Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι πολύ δύσκολο να σεβαστούμε τον νόμο. Συνεπώ, η εργασία η οποία έχει επιτευχθεί είναι πάρα πολύ καλή και βεβαίως ε, έγιναν και τροπολογίε στο κείμενο της Κομισιόν και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω πως λοιπόν η προστιθέμενη αξία είναι πολύ σημαντική για τον ευρωπαϊκό πολίτη. Θα ήθελα να πω ακόμη όσον αφορά την ακόμη περαιτέρω απλοποίηση του κειμένου και τη βελτίωση όσον αφορά τα προγράμματα και την προσβασιμότητα. Έχουμε δει δηλαδή ότι υπάρχουν πράγματα οποία έχουν παρουσιαστεί και ότι πόσο σε ορισμένο βαθμό σε πολλές χώρες υπήρχε μια άχνοια αυτών των θεμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάρτιση, το κείμενο αυτό θα επιτρέψει να ενισχυθεί η διαφάνεια και όπως οι συνάδελφοί μου προφανώς είναι ένας, κανό, ένας αγώνας τον οποίο κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν βεβαίως επιτεύχθη, δεν εστέφθη με επιτυχία, αλλά υπάρχει η αρχή της κοινότητας που λέει ότι η Ένωση στην πολλαπλότητα και στην ιδιαιτερότητα του καθενός και αυτό δίνει τη δυνατότητα, ιδιαίτερα στο γλωσσικό επίπεδο, να χρησιμοποιούνται όλες οι γλώσσες και να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, η ποικιλία. Κάτι άλλο τώρα όσον αφορά την απλοποίηση, φρονώ πως αυτό το οποίο προτείνεται εκ μέρους των συναδέλφων με στήριξη της Κομισιόν όσον αφορά την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την, τις περιοδικές εκθέσεις οι οποίες θα γίνονται. Αυτά όλα θα μας επιτρέψουν να καλύψουμε τις άγνοιες των σωμάτων εκείνων, δικαστικών δικηγόρων κλπ, οι οποίοι δεν γνωρίζουν αυτή τη δυνατότητα την οποία έχουν στα χέρια τους και νομίζω πως αυτό το monitoring, αυτή η παρακολούθηση εκ του σύνεγγης μπορεί να, καλέσει, να καλέσει τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και άλλες χώρες που οι οποίοι αγρούν εντελώς την ύπαρξη αυτής της δυνατότητας. Τρίτη παρατήρηση που θα προσέθετα, η οποία είναι κάτι πολύ γνωστό και παραμενόμενο, ότι δηλαδή ο φάκελος ο οποίος απριόρι φαίνεται πολύ σημαντικός αλλά εκ των προτέρων πολύ σημαντικός αλλά δεν είναι ικανός ότι θα πρέπει να ξέρουμε να θέτουμε τις προτεραιότητες. Δύσκολες εποχές διάγουμε και θα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχουμε θέσει και να βασιστούμε σε προγράμματα εκείνα τα οποία έχουν μία προστιθέμενη αξία, πράγμα το οποίο δίνει μια διάσταση καθαρά ευρωπαϊκή και πιστεύω πως είναι μια αναγκαιότητα για μας. Τελειώνοντας θα επιμείνω σε κάτι ακόμη, κάτι το οποίο ήδη ελέγχθη και εκ μέρους της Κομισιόν και εκ μέρους των συναδέλφων και από τις τροπολογίες ότι θα πρέπει να είναι η κατάρτιση των νομικών, όχι γλωσσικά μόνο, αλλά για μία περαιτέρω εναρμόνιση και την άμεση εφαρμογή των νόμων. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτό τον κοινό ευρωπαϊκό νομικό χώρο εάν δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι συμμετέχοντες, οι παίκτες, οι δράστες σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε πιο σύντομοι γιατί έφτασε στο μεταξύ και ο δεύτερος συγγετής, ο κύριος Μπερλίνγκουερ, και θέλουμε να προλάβουμε να ακούσουμε και τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, της Δανικής Προεδρίας και ο χρόνος τρέχει. Κύριε Μπερλιγκουέρ, μπορείτε να μας κάνετε μια σύντομη ανακεφαλαίωση της ε, γνωμοδότησης ε, της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, και είτε είστε ο συνεισηγητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, είμαι ενόχος. Όχι εντελώς βεβαίως, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά νιώθω πάρα πολύ άσχημα, αλλά όπως να έχουν τα πράγματα πρέπει να πω ότι έχω να πω. Συνεπώς, ο κύριος Κλάης και με αυτόν συνεργαστήκαμε πάρα πολύ με κοινή συνεννόηση και είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συνεδρίαση της κοινή Επιτροπής, να παρουσιάσουμε μια κοινή έκθεση και έχουμε καταμεριστεί τις εργασίες και τις αρμοδιότητες και θα πρέπει να υπογραμμίσω πως βρήκαμε ένα κοινό έδαφος απόλυτης συνεργασίας. έχουμε εξετάσει την πρόταση της Κομισιόν που επακριβώς αφορά το πρόγραμμα δικαιοσύνη 2014-2020. Βεβαίως συνολικά υπήρξε μία σύγκληση σε όλα αυτά τα θέματα προσπαθήσαμε να εισαγάγουμε λομπέρε τροπολογίε βεβαίω σε αυτό το κείμενο, τι οποίε θα τι συνοψίσω πάρα πολύ σύντομα σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε κατά νου. Και είναι και το σημείο εκείνο το οποίο υπογραμμίστηκε μόλι προηγουμένω από την σα και το οποίο αναφέρεται στο πρόγραμμα τη Στοκόλμη. Και φαινόταν ότι πραγματικά με είχε προκαλέσει την προσοχή της Κομισιόν και βέβαια σε αυτό το πρόγραμμα της Στοκόλμης όχι μόνο υπάρχει η δημιουργία ή ευρωπαϊκός χώρος αυτός δικαιοσύνης, δικαϊκός χώρος, αλλά και τη δημιουργία μιας δραστηριότητας η οποία, η οποία θα είναι η βάση για αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν θα δημιουργούσε μια κουλτούρα, μια, ένα πολιτισμό νομικό, αν θέλετε μεταξύ των οποίων θα ήταν δικηγόροι, νομικοί, δικαστές κλπ. οι οποίοι θα περνούσαν από διάφορα στάδια και θα μπορούσαν κατά αυτόν τον τρόπο να φτάσουν να έχουν όλο τον πλούτο και την παράδοση των διαφόρων νομικών καθεστώτων των διαφόρων χωρών πράγμα το οποίο θα ήταν δυνατό να βρεθεί ένα κοινό έδαφος στο οποίο θα μπορούσαν να συνεργαστούν καθώς επίσης και συνεργασία με το Common Law βλέποντας πως πραγματικά είμαι υπέρ αυτής του πράγματος και το δίκαιο δεν είναι μόνο οι δικαστές ε, των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων αλλά είναι και οι εθνικοί δικαστές το δίκαιο βασίζεται σε αυτούς ιδιαίτερους και όχι μόνο Ευρωπαίους δικαστές σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια κατάρτιση μια ε, εκπόνηση καλύτερα μιας νομικής ε, νοοτροπίας παιδείας η οποία, η οποία θα δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτή η παιδεία, αυτή η νοοτροπία η ευρωπαϊκή, ότι υπάρχει και ότι είναι κοινή αυτή και κοινώ αποδεκτή. Καθώς επίσης και η λειτουργία της, η καθημερινότητά της, η καθημερινότητά της. Και νομίζω πως αυτή η εργασία είναι τέτοια και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί συνεργασία σταθερή και μόνιμη μεταξύ των δικαστών η οποία μπορεί να βοηθηθεί πάρα πολύ σε όλες τις τυχές συνεργασίες αυτές που θα μπορούσε να γίνει και οι οποίοι αποτελούν αυτή η συνεργασία δυστυχώ είναι μέχρι στιγμή πάρα πολύ περιορισμένη μεταξύ των δικαστών, μεταξύ των διαφορών χωρών μελών. Αυτό είναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μάζα τεράστια νόμων σε όλη και νομοθετική εργασία. Αυτοί που χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη δεν ξεπερνάνε το 2, 3, 4, 5%. Δεν έχουμε δηλαδή αυτά αποτελέσματα με αυτή την προσπάθεια. Έτσι λοιπόν η δυνατότητα να δημιουργηθεί αυτή η ευρωπαϊκή παιδεία, η νοοτροπία, η νομική αν θέλετε, είναι ότι υπέρα απαραίτητο για να χρησιμοποιηθεί υπέρα απαραίτητο, διότι πραγματική γίνεται όλη αυτή η νομοθεσία, αλλά για ποιο να γίνεται αυτή η νομοθεσία, αυτό το νομοθετικό έργο λοιπόν. Έτσι λοιπόν Όλα αυτά τα πράγματα θα τα δείτε γραμμένα μέσα στη δική μου έκθεση και θα δείτε και μια σειρά όλων μέτρων για τη δυνατότητα αύξησης ε, της κατάρτισης, όπως, όχι όπως παλαιότερα που γινόταν μέσα των σχολών, αλλά νέες μορφές συνεργασίας, ε, ένταξης, ενσωμάτωσης, ξεκινώντας από συγκεκριμένες περιπτώσεις, δίνοντας την εμπειρία την οποία χρειάζεται ο καθένας για την δική του άσκηση του επαγγέλματος στα πλαίσια του δικού του δικαστηρίου, στα πλαίσια της δικής του ε, δικαστικής απασχόλησης κατά αυτόν τον τρόπο να υπάρχουν ανταλλαγές άμεσες, όχι μόνο πηγαίνοντας δικαστές από εδώ, εκεί και λοιπά, από ένα δικαστήριο στο άλλο, στο οποίο μπορεί να γίνει πραγματικά, αλλά με πολύ λίγο μικρό αριθμό, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Ζητάμε κάτι περισσότερο, εμπειρία, πολύ μεγάλη εμπειρία, την οποία μπορούμε να μεταφέρουμε για να, για παράδειγμα έχουμε οι Ολλανδοί, δημιουργούσαν στα δικαστήρια, σε κάθε δικαστήριο, έναν ρεφεραντέρ, έναν ε, αναφερόμενο στα θέματα αυτά, ο οποίος ασχολείται ειδικά με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Και βεβαίως υπάρχει ένα κέντρο, ε, ένα κέντρο μορφωτικό θα λέγαμε, το δικαστικό μορφωτικό, το οποίο ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Οι Ολλανδοί υπήρξαν λοιπόν οι πρωτοπόροι σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπελίνγκουαλ. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε και την κυρία Γκόνση της και η γητριά μας. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλει να προσθέσει κάτι, και στους υπόλοιπους φυσικά. Η κυρία Γκόντς, θα είμαι επιγραμματική γιατί καλύφθηκαν τα περισσότερα ουσιώδη ζητήματα από τους συνεισηγητές. Είμαι βεβαία ότι η έκθεση θα είναι καταπληκτική και στη συζήτηση με τη Δανική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πράγματα ήταν πολύ θετικά. Οι προετοιμασίες βαίνουν καλώς λοιπόν. Αναφέρθηκε η αποδοχή της απλούστευσης της διαδικασίας και η ελάφρυνση του διοικητικού άχθους για τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που επίσης ε, υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση κονδυλίων. Ε, Επίση ε, είπαμε ελαστικότητα, προβλεψιμότητα και διαφάνεια. Όλες αυτές οι έννοιες είναι σημαντικές, γι' αυτό ε, είπαμε μέσω και των κατεξουδάτσι πράξεων και παρά από αυτές να έχουμε και εμείς κάποιο λόγο ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, συνοχή, συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα και άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς. Πολύ σημαντικό είναι να έχουμε συγκεκριμένους και σωστούς δείκτες. Και καλό θα ήταν να τους έχουμε ήδη από την αρχή της διαδικασίας. Συζητήθηκε το κατά πόσο θα πρέπει να κατονομάσουμε κάποια πανευρωπαϊκά δίκτυα. Μετά συμφωνήσαμε ότι αυτοί που δεν αναφέρονται στα άρθρα να αρχίσουμε να κατανομάζουμε συγκεκριμένα δίκτυα είναι σαν να αποκλείουμε μερικούς. Προτιμώ να αφήνουμε ανοιχτό το θέμα αυτό. Αναφέρονται ενδεικτικά στις αιτιολογικές σκέψεις κάποια παραδείγματα. Το θέμα του κράτους δικαίου και η δικαστική εξουσία σε ένα δημοκρατικό σύστημα είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης η ενημέρωση για το κοινοτικό δίκαιο και η ενημέρωση για τα δικαιώματα, πολύ σημαντικά θέματα. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις, τις δικαστικές πρακτικές, να επενδύσουμε στην παιδεία, στην ε, ενημέρωση των εισαγγελέων, των δικαστών, αλλά να αφιπλήσουμε και το κοινό ε, Ω προ τι διακρίσει. Επίση, ίση πρόσβαση, ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ιδιαίτερα για του πιο ευάλωτους συμπολίτε μα οι σχετικές τροπολογίες και φαίνεται ότι θα περιληφθούν στην τελική πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Γκέντς. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο, αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι, γιατί ήδη έχουμε εξαντλήσει το χρόνο μας. Καλώς. Θα είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι για την έκθεση και για την αγαστή συνεργασία που είχαμε και με τη Δανική Προεδρία και με τους συνεισηγητές. Άκουσα σήμερα πολλές ιδέες και προτάσεις και μερικές από αυτές ήδη περιλαμβάνονται στην έκθεση. Για το θέμα της κατάρτισης των δικαστών και των ονομαθών Πιστεύουμε ότι το θέμα της επιμόρφωσης, της κατάρτισης ε, έχει νευραλική σημασία σε αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης που θέλουμε να διαμορφώσουμε και να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη. Άκουσα βέβαια και άλλες έννοιες όπως τη διαφάνεια, την απλούστευση, την παρακολούθηση, τους δείκτες, την ε, χρήση, ε, αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών και πιστεύω ότι με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμπλουτισμένη με τις τροπολογίες θα καταλήξουμε στον κοινό μας στόχο. Έχουμε βέβαια κάποιες επιφυλάξεις και ανησυχίες για ορισμένες τροπολογίες που αφορούν την εφαρμογή. Γιατί πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της προστιθέμενης αξίας, της απλούστευσης αλλά δεν θα πρέπει ταυτόχρονα να δημιουργούμε περί το άχθος και να επιβαρύνουμε αυτή τη διαδικασία χωρίς λόγο. Επίσης θέλουμε να πετύχουμε εμπρόθεσμη εφαρμογή του σχεδίων, ιδιαίτερα για τους δικαιούχους, προς δικό τους όφελος. Γιατί αυτό είναι το αίτημα που ακούμε συνεχώς. Ότι με το νέο αυτό σχέδιο θα πρέπει να βελτιώσουμε τις προηγούμενές μας αδυναμίες και τα κενά του, των προηγούμενων προγραμμάτων. Και αυτό είναι και το ζητούμενο. Πάντως ε, είμαι βεβαία ότι θα καταλήξουμε σε πολύ αισιοπέρας και θα βρούμε τα κατάλληλα προγράμματα που θα ανταποκρίνονται στον κοινό μας στόχο και επιθυμία. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο τώρα μήπως θα ήθελε να πει δύο λόγια. Σύντομα παρακαλώ. Η κυρία Γκάρτ. Νόρινγκ λέγομαι. Καλώς, θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι λακωνική. Όπως ξέρετε το Συμβούλιο πρόσφατα είχε στις 8 Ιουνίου το Συμβούλιο Τζάι και ε, συμφώνησε για μια μερική και γενική προσέγγιση του προγράμματος για τη δικαιοσύνη. Η γενική προσέγγιση καλύπτει το σύνολο του προγράμματος πλην του προπολογισμού που θα γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευση σε άλλο Υπουργικό Συμβούλιο. Χαιρόμαστε για ότι το σχέδιο έκθεσης ε, ευθυγραμμίζεται με τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, κάτι που θα διευκολύνει τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις ε, μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Γνωρίζω ότι ε, και οι συνεισηγητές και το Συμβούλιο συμφωνούν με το στόχο της πρότασης, δηλαδή θέλουμε μια απλουστευμένη και συνεκτική προσέγγιση για να αναπτύξουμε καλύτερα τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης οι συνεισηγητέ για το Συμβούλιο ευθυγραμμίζονται σε πολλά κέρια ζητήματα. Για παράδειγμα, συμφωνούμε ότι οι χρηματοδοτούμενε δράσει θα πρέπει να αποδεικνύουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του και να υπάρχει σαφή σαφής ορισμός της έννοιας αυτής στο κείμενο. Επίση, συμφωνούμε για του συγκεκριμένου στόχου τη πρόταση να βελτιώσουμε δηλαδή τη δικαστική συνεργασία, να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και επίσης να στηρίξουμε την ε, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστών. Επίση, θέλουμε να συμπεριληφθούν συγκεκριμένοι δείκτε στο κείμενο για να αποτελέσουν τη βάση της διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγηση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα ο χρόνος, στο θέμα του, του συγχρονισμού είναι πολύ κέριο, γιατί το υπάρχον ε, πρόγραμμα ε, λίγη το 2013, οπότε το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα πρέπει να εγκριθεί εγκαίρως. Γι' αυτό και η Ιδανική Προεδρία έχει θέσει ως προτεραιότητα το ζήτημα αυτό στο Συμβούλιο και είχε και άτυπες πολύ επικοδομητικές συναντήσεις με τους συνεισηγητές. Έτσι πιστεύουμε ότι θα ε, προλιαθεί το έδαφος για συμφωνία το συντομότερο δυνατό μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Τώρα, μήπως θα ήθελαν οι δύο συνεισηγητές να πούν το τελικό λόγο. Γιατί ακούσαμε το Συμβούλιο, ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει κάποιος από τους δύο εισηγητές να ανακεφαλαιώσει. Ο κύριος Κλέης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν του ηγητέ μα, του κύριο Φίνιπα και κύριο Κούνκετ, οι οποίοι είναι οι σκιώδει Νομίζω πως φαίνεται αυτή τη στιγμή πως υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση όσον αφορά τη ρεκπόληση αυτή τη έκθεση. Δεν θα περάσω αυτή τη στιγμή στι λεπτομέρειε όλε, αλλά έχω την εντύπωση ότι με ένα γενικό τρόπο είμαστε όλοι προ την αυτή κατεύθυνση, περισσότερη διαφάνεια, απλοποίηση έχουμε δείκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ σαφείς, πράγμα το οποίο μας κάνει να μπορούμε να φτάσουμε στους στόχους που έχουμε θέσει. Η Κομισιόν εξεφράστη όσον αφορά της κατεξουσιοδότηση πράξης. Εδώ θα πρέπει να δούμε τώρα εμείς τι θα αποφασίσουμε επί του πρακτέου, κατά πόσον δηλαδή θέλουμε να δεχθούμε αυτές τις κατεντοεξουσιοδότηση πράξεις ε, δίνοντας ενταυτό στο, δικαστή, στο κοινοβούλιο συγγνώμη, τη δυνατότητα για τη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων τις οποίες έχουμε θέσει. Πράγμα το οποίο βεβαίως δεν θα αποτελέσει ένα χάσιμο χρόνου διότι μπορεί να γίνει μια καλή συνεργασία μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου, διότι βρισκόμαστε στην, αυτή, στην ίδια γραμμή Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι περίπλοκα και ότι θα πάνε όλα τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ ο Πρόεδρο. Φρονώ πως περατώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο την έκθεση αυτή, πράγμα το οποίο μας επιτρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους συμμετέχοντας σε αυτή τη κυρία συζήτηση μεταξύ της Νομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ελευθεριών και θα περάσουμε τώρα στο θέμα δίκαιο και ηθαγένεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, ιδιαίτερα την κυρία Ισηγήτρα για την παρουσία της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λαμπρά. Προχωρούμε. Στο επόμενο θέμα, δικαιώματα και ηθαγένεια, πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020. Θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεση τη κυρία Γκέντς και θα καθορίσουμε και την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Η συγκεκριά μα για το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια είναι η συνάδελφο Κίνγκα Γκέντ. Θα μα παρουσιάσει λοιπόν το σχέδιο έκθεση για το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια, Δάφνη 3 και ενότητε πολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία και ισότητα των φύλων του προγράμματο Απασχόληση και Κοινωνική Αλληλεγγύη Progress. Τα προγράμματα αυτά εμπίπτουν εν μέρη στις αρμοδιότητες και άλλων επιτροπών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Επιτροπής Γυναικών, με βάση τον ε, διαδικαστικό κανόνα 50. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα την εισηγήτρια, μετά τη Δανική Προεδρία και κατόπιν θα γίνει συζήτηση. Κυρία Γκέντς, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια είναι παρόμοιο με το προηγούμενο που συζητήσαμε. Και οι ανησυχίες και το μέλημα είναι παρόμοιο. Δηλαδή, έχουμε συγχώνευση των τριών προγραμμάτων, των προγραμμάτων Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια, Δάφνη 3 και την καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία και ισότητα των φύλων, ε, του προγράμματο Απασχόληση και Κοινωνική Ελληνική, αυτά τα τρία προγράμματα συγχωνεύονται πια και μετατρέπονται σε ένα πρόγραμμα Δικαιώματα και ηθαγένεια. Εμεί προτείνουμε αλλαγή του προγράμματο ε, από το δικαιώματα και ηθαγένεια στο δικαιώματα ισότητα και ηθαγένεια, γιατί νομίζω ότι έτσι αντανακλούμε καλύτερα το πραγματικό, το ουσιαστικό περιεχόμενο του προγράμματο και δίνουμε και καλύτερη έμφαση στα επιμέρους του στοιχεία, γιατί Είχαμε πολλέ διαβουλεύσει και με εκπροσώπου κοινωνία των πολιτών, με την Επιτροπή, με τη Δανική Προεδρία, η οποία δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα ξεκινώντα από νωρί άτυπο τριμερή διάλογο για το θέμα αυτό. Οπότε έχω την εντύπωση ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο και με τη Δανική Προεδρία και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε στα πιο σημαντικά θέματα. Δημιουργήθηκε ήδη μια πολύ καλή βάση και φυσικά συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Βέβαια, ε, αυτό που με στεναχωρεί κάπως είναι η αναδιάρθρωση των κονδυλίων μετά τη συγχώνευση των ε, τριών προγραμμάτων, κάτι που οδήγησε σε μείωση του προγράμματος ε, ισότητα των φύλων με την αναδιάρθρωση των κονδυλίων το προτινόμενο ποσό είναι μικρότερο από, τα, από το άθροισμα των ε, τριών προηγούμενων. Γιατί λοιπόν ε, μείωσε το ποσό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς ε, θέλαμε έστω και μία μικρή αύξηση, όχι όμως μείωση. Βέβαια, με την κρίση βλέπουμε όλο και περισσότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κρίμα ε, το μέλημά μας για την προστασία τους να μην αντικατοπτρίζεται σε έναν πιο ενισχυμένο προϋπολογισμό. Επίσης, ε, η ελαστικότητα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για το μέλλον, αλλά αυτό που για μας είναι το πιο σημαντικό είναι το πρόγραμμα να έχει κάποια προβλεψιμότητα για τους ετούντες ε, τα κονδύλια. Και επίσης θα πρέπει να γίνεται ε, μια σαφής κατανομή και ισότιμη κατανομή στο ετήσιο πρόγραμμα μεταξύ των διαφόρων στόχων. Θα πρέπει λοιπόν να, ε, να συμφωνήσουμε και να επηρεάσουμε ε, και εμείς την επιλογή των προγραμμάτων. Γι' αυτό και μετά από μακροχρόνια συζήτηση καταλήξαμε και πάλι στη μέθοδο των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Απλούστευση σημαίνει και ευκολότερη εφαρμογή και διαδικασία αναφορά των ετούντων. Έχουμε μια άρση λοιπόν, η ελάφρυνση του διοικητικού άχθους, όπως και στο πρόγραμμα δικαιοσύνη. Επίσης το θέμα της γεωγραφικής, ισόρροπης γεωγραφικής κατανομής είναι πολύ σημαντικό, καθώς και της ε, αρρωγής προς τα κράτη-μέλη που δεν υποβάλλουν καθόλου αιτήσει για μερικά χρόνια. Και πάλι είχαμε το δίλημα να αναφέρουμε ή να μην αναφέρουμε συγκεκριμένα ονόματα δικαιούχων ε, ευρωπαϊκών δηλαδή δικτύων που ήταν δικαιούχοι στα προηγούμενα προγράμματα. Τελικά αποφασίσαμε να μην ονοματίσουμε συγκεκριμένους ε, οργανισμούς, απλώς να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που θα είναι αρκετά ευρύ, αλλά και αρκετά συγκεκριμένο, ώστε να καλύπτει τα πιο σημαντικά δίκτυα. Άλλο σημαντικό θέμα είναι να υπάρχει με συμπληρωματικότητα και συνοχή του προγράμματος αυτού με άλλα προγράμματα και με το έργο άλλων ε, κοινοτικών οργανισμών όπως ε, του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα με τον οποίο είχαμε συζήτηση χθες. Επίσης, δεν θα πρέπει να, σε, να το πεδίο εφαρμογή ε, ε, υπερβολικά ε, πέραν των ε, ιδιωτών, αλλά είπαμε να περιληφθούν και η πήκοοι τρίτο χωρών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το θέμα των, της συμμετοχής μας σε διεθνείς συμβάσεις θα πρέπει να αναφέρεται στο πρόγραμμα. Επίσης αναφέρεται το πρόγραμμα ισότητα για όλους, ειδική μνήμα και επίσης ειδική μνήμα της καταπολέμησης των διακρίσεων. Πολύ σημαντικό στους χαλεπούς καιρούς της κρίσης που διανύουμε. Επίσης έχουμε μια διαβρύση των στόχων, καταπολέμηση της, α, της μυσαλλοδοξίας, της εξύμνησης ε, του μίσους. Επίσης, ε, καταδικάζουμε την βία κατά των γυναικών, παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων. Προστατεύουμε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Θέλουμε και εθνικά προγράμματα, αλλά και προγράμματα μικρής κλίμακος, που θα έχουν ευρωπαϊκή όμως προστιθέμενη αξία. Επίσης θέλουμε ορατότητα, προβολή των προγραμμάτων μεταξύ των ετούντων, ειδικού δείκτες, το συντομότερο δυνατό. Να ευχαριστήσω λοιπόν και τη Δανική Προεδρία για τη μέχρι τώρα πολύ επικοδομητική συνεργασία που ελπίζω ότι θα συνεχιστεί. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Γκάντς. Να ακούσουμε πάλι την Επιτροπή, το Συμβούλιο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ καλωσορίζω για άλλη μια φορά τη συνεργασία μας, το σχέδιο έκθεσης αυτό. Θεωρούμε ότι είναι μια εξαιρετική βάση για τα επόμενα βήματα της συζήτησης. Συμφωνούμε ότι υπάρχουν εδώ πιο σαφείς στόχοι, πιο καλά παρουσιασμένοι. Και θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα, γιατί μειώθηκε ο προϋπολογισμός, ερώτηση της εισηγήτριας. Θεωρούμε ότι σήμερα υπάρχει μία ευελιξία μεταξύ αυτού του προγράμματος και άλλων προγραμμάτων, κάτι που μας επιτρέπει να καθορίσουμε τις δράσεις. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι κάποιες δράσεις θα παραμείνουν χωρίς χρηματοδότηση. Θέλω επίσης να πω ότι τελικά θα συμφωνηθεί το πρόγραμμα αυτό από τους νομοθέτες και πρέπει σε κάθε περίπτωση να εγγυηθούμε αυτήν την απλοποίηση, τη διαφάνεια και βεβαίως συμφωνούμε και με την γεωγραφική κατανομή και κάλυψη αλλά σαφώς και θα πρέπει να δοθεί στους δικαιούχους δυνατότητα για στοχευμένες δράσεις. Σε καμία περίπτωση ε, δεν θέλουμε κάτι διαφορετικό από το Κοινοβούλιο, δηλαδή αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων. Το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Συμβούλιο συμφώνησε για μια γενική προσέγγιση όσον αφορά το θέμα αυτό δικαιώματα και ηθαγένεια, καθώς και το πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη, που καλύπτει το όλο φάσμα των προτάσεων εκτός ε, από τις πτυχές αυτές που διαπραγματεύονται κάπου αλλού στο Συμβούλιο οι υπηρεσίες μας. Πρόκειται λοιπόν για μια πρόταση που συμβαδίζει με αυτά που εμείς ε, πρεσβεύουμε και βεβαίως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου θα συνεχιστούν στη βάση αυτή. Θα συμφωνήσουμε με την εισηγήτρια ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μια γενικότερη και πιο απλή πρόταση χρηματοδότησης όπως ορίζεται και στο χαρτί μελιωδών δικαιωμάτων και όπως ορίζει και η συνθήκη. Σε πολλά σημεία λοιπόν το Συμβούλιο και η Συγήτρια συμφωνούν. Πρώτον, συμφωνούμε και οι δύο ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να βασίζεται στην απόδειξη της προστιθέμενης αξίας για την Ευρώπη. Δεύτερον, συμφωνούμε ότι ο κατάλογος των πολύ συγκεκριμένων στόχων των προγραμμάτων θα πρέπει να συμπληρωθεί, έτσι ώστε να καλυφθούν σημεία όπως η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός και η συμμεταχείριση βεβαίως ανδρών και γυναικών. Τα προγράμματα αυτά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίσουν και να εγγυηθούν μια ίση κατανομή των πόρων γεωγραφικά αλλά και ανακατηγορίες προγραμμάτων και βεβαίως συμφωνούμε ότι χρειάζεται παρακολούθηση όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων στις διάφορες φάσεις τους. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και αποτελεί ένα από τα σημεία διαπραγμάτευσης. Στο τέλος του 2013 τελειώνει η παρούσα φάση χρηματοδότησης και γι' αυτό το λόγο η Προεδρία της Δανίας θεωρεί προτεραιότητα την συνέχιση αυτών των διαπραγματεύσεων και μέχρι τώρα ήμασταν πάρα πολύ ε, ικανοποιημένοι από τις ανεπίσημες επαφές που είχαμε με την εισηγήτρια. Ήταν εξαιρετικά επικοδομητικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε λίγο χρόνο για συζήτηση. Ο κύριος Μισελ θέλει να πάρει το λόγο. Έχετε το λόγο, κύριε Μισελ. Να συγχαρώ την κυρία Γκένς που έκανε την έκθεση αυτή στηρίζω σε μεγάλο βαθμό τις προτάσεις της και έχω μία μόνο παρατήρηση η οποία μπορεί να σας φανεί ίσως όχι τόσο ουσιαστική. Πουθενά δεν βλέπω, πουθενά δεν βλέπω να γίνεται αναφορά για την βία, μια ιδιαίτερη βία η οποία πολλές φορές ε, είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν αναφέρεται ρητά. Ε, αναφέρομαι στη βία κατά των ηλικιωμένων, στο εσωτερικό των οικογενειών, αλλά όχι μόνο. Και θέλω να καταθέσω μια τροπολογία έτσι ώστε να αναφέρουμε ρητά αυτήν την βία. Δεν είναι μια κλασική βία, είναι μια βία κατά κάποιο τρόπο κρυμμένη. Κανείς δεν ε, τολμάει να αναφέρει αυτήν την βία. Υπάρχει όμως παρόλα αυτά και κάπως θα πρέπει να το καλύψουμε με μια ειδική τροπολογία. Θέλω λοιπόν να καταθέσω μια τροπολογία για το συγκεκριμένο αυτό θέμα και όπως ξέρετε οργανώνουμε και ένα φόρουμ με ειδικού, με μάρτυρες και τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται στο εσωτερικό των οικογενειών. Κατά τα άλλα, βεβαίως και στηρίζω τις τροπολογίες της ηγήτριας. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόγκς. Uh, Ευχαριστώ. Η ηθαγένεια είναι μια ψεύτικη νόημα γιατί πραγματικά υπάρχουν υποχρεώσεις οι οποίες ε, προκύπτουν από την εθνικότητα και αυτό κατά τον στην Ευρωπαϊκή, στην Ανατολική Ευρώπη κατοκαταλαβαίνει το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι θέλω να πω, αλλά δείτε υπάρχει πραγματικά μια σύγχυση. Η ηθαγένεια πρέπει να βασίζεται στην εθνικότητα και διαφορετικά υπάρχει η διάκριση η οποία γίνεται. Νομίζω πως είναι πολύ πολύ σημαντικό στα πλαίσια της δημοκρατίας, δημοκρατία όπου ο λαός πραγματικά είναι κυρίαρχος και τώρα αποτελεί κανένας μέλος του έθνου δεν σημαίνει πραγματικά ότι δεν σημαίνει ότι μπορεί να εκλέγει οποιονδήποτε, πράγμα το οποίο θα, δημιουργεί το χάος. Έτσι λοιπόν το θέμα της ε, ηθαγένειας μπορεί να αναφέρεται και σε πολίτες τρίτες πολίτες. Ποια είναι αυτή τα δικαιώματα. Υπάρχουν πολλές ειδών που υπάρχουν ε, ποιες είναι οι δυνατότητες οι οποίες δίνονται σε αυτά. Βεβαίως κάθε κάθε άνθρωπος θα πρέπει να προστατεύεται ανεξάρτητα στα γενία του και της προέλευσής του. Βεβαίω θα πρέπει να έχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να έχει ένα επάγγελμα, να υπάρχει και όλες εκείνες τις κοινωνικές παροχές. Ωστόσο, αν τώρα διευρύνουμε πάρα πολύ αυτό αυτόν τον όρο, δεν ξέρουμε πραγματικά πού βρίσκεται η θα γίνει αν βάλουμε όλα αυτά στη μέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος Συγγνώμη πάρα πολύ ότι δεν μπόρεσα να εργαστώ επί της εκθέσεως αυτής πάρα πολύ. Ένα πράγμα όμω που με ανησυχεί πάρα πολύ και θα καταθέσω τροπολογίες από το θέμα αυτό. Η ηθαγένεια είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο πρόγραμμα αυτό. Εργαστήκαμε στα εμπόδια της ηθαγένειας τα οποία υπάρχουν σε μια έκθεση που κάναμε πρόσφατα. Τώρα εργαζόμαστε χώρο πολύ περισσότερο στους πολίτες και τη, την πολιτική ταγένεια, τη σχετισμό και βρισκόμαστε σε μια ηθαγένεια παθητική θα έλεγα, δηλαδή πώς θα αναγνωρίσουμε τα δικαιώματα αλλά η ηθαγένεια σε αυτά, τα πλαίσια αυτού εδώ του σώματος θα πρέπει να θεωρηθεί περισσότερο σε μια ενεργός και όχι παθητική έννοια. Δηλαδή ο πολίτης θα πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία την αποφασιστική διαδικασία και των αποφάσεων. Αυτό το στοιχείο λοιπόν είναι αυτό το οποίο είναι απόν από το κείμενο αναχείρας και μου φαίνεται πως υπάρχει μια ανάγκη να εργαστούμε πολύ περισσότερο με το πρόγραμμα Ευρώπη των Πολιτών που είναι προγράμματα παράλληλα και όπου μου φαίνεται ότι υπάρχει και η Επιτροπή Παιδείας η οποία εργάζεται για αυτά τα θέματα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει κάποια συνεργασία. Υπό την επιφύλαξη ότι θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα πράγματα θα πρέπει να ειδωθούν, σας τα υποβάλλω όλα αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πριν επανέλθω στον εισηγητή, δεν βλέπω άλλα χέρια. Α, η Κομισιόν μήπως θα ήθελε να, να πει δύο λόγια παρακαλώ. Κύριε Μίχου, πιστεύω πως το πρόγραμμα μόλις αναφέρθηκε και θα ήθελα να το διευκρινίσω για να υπάρχει σύγχυση. υπάρχουν ένα πρόγραμμα για την ηθαγένεια ε, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας. Όλα αυτά τα σχόλια λοιπόν τα οποία έχουν γίνει καθώς και αυτό το σημείο ότι μπορούν να συμπεριληφθούν. Το πρόγραμμά μας λοιπόν που έχουμε αυτή τη στιγμή αναχείρας ε, για παράδειγμα, προσπαθούμε να έχουμε μια συνοχή με τα διαφόρων των project και τα διαφόρων προγραμμάτων σχεδίων που έχουμε και το τελευταίο ε, σχόλιο το οποίο είχα είναι περισσότερο για αυτό το σχέδιο όσον αφορά την επικοινωνία, την ανακοίνωση. Εκεί θα μπει περισσότερο παρά στο παρόν. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια δεν υπάρχουν ούτε από την Προεδρία, οπότε κύριε Γκέντς έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους όσους ε, έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Ήταν σαφές ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματος και με την Προεδρία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο, ο κύριος Λουί Μισελ μίλησε για τη βία κατά των ηλικιωμένων. Περιμένω τι τροπολογίες του, πολύ ευχαρίστω για να το συμπεριλάβω. Πάντα αντιμετωπίζουμε το δίλημα ότι αν αρχίσουμε και κάνουμε κατάλογο όλων των ευάλωτων ομάδων διατρέχουμε τον κίνδυνο ξεχάσουμε μερικούς. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες ευάλωτες ομάδες, αλλά δεν είναι εξαντλητική η αναφορά. Πάντως συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μισελ ότι είναι σημαντικό πρόβλημα, υπάρχει, αλλά δυστυχώς ε, μιλούμε πολύ λιγότερο για την βία κατά των ε, ηλικιωμένων παρά για τη βία κατά των ε, γυναικών, παιδιών κτλ. Κύριε Μπρόνς, είπαμε να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή και στους υπηκούς τρίτων χωρών που είτε είναι αιτούντες άσυλο είτε διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μετανάστες, αποσπασμένοι κτλ. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να εγγυηθούμε τα δικαιώματα και των ανθρώπων αυτών, που δεν είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά διαμένως αυτοί. αυτή. Υπάρχει και το θέμα του τι θα καλύψουμε από το συγκεκριμένο ταμείο και τι δραστηριότητες θα καλυφθούν από άλλα ταμεία. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια συνοχή και συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων. Πάντως συμφωνώ ότι η ηθαγένεια δεν θα πρέπει να είναι μόνο παθητική αλλά και ενεργητική το ενεργητικό σκέλος είναι πολύ σημαντικό. Θα δούμε πώς θα το περιλάβουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η 5η Ιουλίου είναι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Έχουμε λίγο χρόνο, περιμένω τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ. Ακριβώς εμείς σας ευχαριστούμε κυρία Γκόντς, ειδικά για την τελευταία σας παρατήρηση, για τη διορία για τις προθεσμίες, για τις ε, τροπολογίες, συγγνώμη. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι τροπολογίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 5 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Και το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση είναι το εξή. Εξέταση των τροπολογιών στην Επιτροπή μας στις 19 Σεπτεμβρίου και ψηφοφορία προς ανατολισμού στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και πάλι θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου. Τα σημειώσατε όλα αυτά που σας είπα. Πολύ ωραία, άλλα σχόλια δεν υπάρχουν. Οπότε... Το επόμενο σημείο έχει προγραμματιστεί για τις 10.30. Η συγγετρία είναι η κυρία Χολμάιερ. Δεν έχει έρθει ακόμη. Οπότε προτείνω σπάνιο για την Επιτροπή μας να κάνουμε ένα 20 λεπτό διάλειμμα Εν αναμονή τη κυρία Χολμάιερ, γιατί το δικό τη θέμα, επαναλαμβάνω, προγραμματίστηκε για τι 10.30 και θα μα υποβάλει την ενδιάμεση έκθεση σε ό,τι αφορά την αίσια έκβαση των διαπραγματεύσεων για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Οπότε, 10 και μισή παρακαλώ να επιστρέψετε στην αίθουσα για να συνεχίσουμε.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 colleagues, as we foresaw, our colleague Mrs. Holmeyer is already here to present the draft opinion on the interim report on... Για να παρουσιάσει την έκθεση της κυρίας συνάδελφας, όχι. έκθεση και το 2014-2020 παρουσιάζουμε την έκθεση της Επιτροπής για το πρόγραμμα το οποίο αφορά αυτή την περίοδο. Το τα διάφορα προγράμματα τα οποία το περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα Περικλής. και ε, έκθεση εν ώψη θετική έκθεση διαδικασία έγκριση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Πρόεδρε, βλέπω ότι πάρα πολλοί βουλευτές είναι εδώ σήμερα, άρα είμαστε μεταξύ μας και άρα μπορούμε να συζητήσουμε για το πρόγραμμα το πολιετές 14-20, 2014-2020. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την εξαιρετική συνάντηση που είχαμε μεταξύ των εισηγητών Ξέρετε ότι για μια γνωμοδότηση δεν μπορούμε σε μια σελίδα και ούτε μια σελίδα να βάλουμε όλα αυτά που θα θέλαμε να βάλουμε, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πραγματικά ακούστηκαν ε, οι προτάσεις των ΜΕΝ και των ΔΕ και μπορέσαμε να έχουμε μια πάρα πολύ επικοδομητική συνεργασία. Τώρα, όσον αφορά τη διάρθρωση αυτής της ε, πρότασης, Είχα διάφορες προκαταρτικές ε, συζητήσεις και είχα πει ότι δεν έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά γιατί η ασφάλεια των τροφίμων μπαίνει μέσα στο θέμα της ασφάλειας των ε, πολιτών και το θέμα της δικαιοσύνης. Δεν κατάλαβα γιατί αυτά όλα εμπεριέχονται στην ίδια κατηγορία. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να ζητήσουμε ε, κάποιες διευκρινήσεις και αυτό το έχω αναφέρει στην γνωμοδότηση. Δεύτερον, και εδώ βεβαίως πάντα θα μιλήσω για τη διάρθρωση των κονδυλίων, των πόρων. Ένα μεγάλο τμήμα αυτών προέρχεται από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε για το νομικό κομμάτι και έχω την εντύπωση ότι αυτό τελικά είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής ε, Γιούρη. Εκεί πρέπει να μπει η έμφαση, αν θέλετε. Εκεί έχει μπει η έμφαση. Και πάλι όσον αφορά τη διάρθρωση των πόρων, θα ήθελα να πω ότι αυτή η αναδιάρθρωση είναι θετική, επιτυχής θα έλεγα, και ότι ουσιαστικά υπάρχουν ε, διάφορες διευθετήσεις για οριζόντια διευθέτηση και διοίκηση και μου φαίνεται ότι επικράτησε η λογική. Βεβαίως πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες για να δούμε πιο ειδικά τι ε, είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά σε γενικές γραμμές πραγματικά επικράτησε η λογική. Για τη μετανάστευση, για τη μετανάστευση θα ήθελα να πω ότι βεβαίως μπορεί κανείς να πει ότι το θέμα εξαρτάται, αν δηλαδή είναι αρκετά ή όχι αρκετά αυτά τα κονδύλια, από τον αριθμό των μεταναστών και από τον αριθμό των ετούντων άσυλο. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό για την συνάδελφό μας την κυρία Γκυγιόμ είναι το θέμα της προστιθέμενης αξίας αυτών των δράσεων σε, ε, για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρουμε ότι υπάρχει το εθνικό σύστημα της κάθε χώρας για την αντιμετώπιση των ετούντων άσυλο. Το θέμα είναι αν αυτά που κάνουμε εμείς εδώ είναι μια προστιθέμενη αξία για τους πρόσφυγες αυτούς καθεαυτούς και όχι απλώς να γίνονται εξοικονομήσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς και περικοπές στα εθνικά προβλήματα. Γιατί ξέρετε ότι οι χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα θέματα αυτά της μετανάστευσης και της ε, παροχής ασύλου είναι χώρες τις οποίες θέλουμε να στηρίξουμε. Τώρα, αυτό που βλέπω σαν ιδιαίτερο πρόβλημα για το ESF είναι ότι αν κοιτάξει κανείς τον προπολογισμό ιδιαίτερα για το 13 βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτά τα εκατομμύρια περικοπές και αν μπούμε στις λεπτομέρειες γιατί δεν δόθηκαν αυτά τα εκατομμύρια, ποιοι είναι οι λόγοι, πώς αιτιολογείται. Ήταν λανθασμένο ο προσανατολισμός του προγράμματος του συγκεκριμένου ή δεν μπόρεσαν να απορροφηθούν κάποια κονδύλια για άλλους λόγους. Διαπιστώνω πάντως ότι αυτά τα 64 εκατομμύρια μείων επαναλαμβάνεται αυτή η μείωση και το 14. Δηλαδή μείων 70 εκατομμύρια βλέπουμε εκεί τώρα όσον αφορά το PNR και την στήριξη που πρέπει να δοθεί σε κάποια κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και αδυναμίες. Τι γίνεται με τη στήριξη της Frontex, επίσης το κέντρο εγκληματικότητας για το άσυλο, Crime Asylum Center. Σε γενικές γραμμές εδώ βλέπουμε ότι χάνεται περίπου το 10% των ε, κονδυλίων της χρηματοδότησης. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και σε μια τέτοια χρηματοδότηση πολυετή, δεν μπορεί κανείς να διαπιστώσει με ξεκάθαρο τρόπο πού υπάρχουν οι απώλειες και ότι πολλές φορές δεν υπάρχει σχεδιασμός, αν θέλετε, χρηματοδότησης. Όταν δηλαδή κάνουμε ερωτήσεις συγκεκριμένες στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνουμε ότι παραδείγματο χάρη μεγάλοι οργανισμοί όπως η Europol για το τμήμα παραδείγματο χάρη της παιδικής πορνογραφίας έχει μόνο πέντε άτομα αρμόδια. Στις Ηνωμένε Πολιτείε. αν συγκρίνουμε τους αριθμούς, είμαστε σε τρομερά μειονεκτική θέση. Για πολύ ευαίσθητα, θέλετε, θέματα, όπως αυτό της παιδικής πορνογραφίας, διαπιστώνουμε ότι στην Ευρώπη ακόμα λείπει προσωπικό, λείπει σχεδιασμός, λείπει πρόβλεψη και γι' αυτό και για τις διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες και την ΕΑΖΟ, για την Europol, για τους διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και υπηρεσίες που παίζουν ένα καθοριστικό δεν υπάρχει η απαραίτητη πρόβλεψη και ανταπόκριση όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Προσπάθησα λοιπόν να λάβω υπόψη όλες τις προτάσεις των συναδέλφων, αλλά σε γενικές γραμμές επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι επικράτησε η λογική και ότι <coughs> τα σημεία τα οποία είχε εντοπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν κέρια σημεία, σαν κεντρικά σημεία, ελήφθησαν υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Χολμάγερ. Try Δυστυχώς ε, το Συμβούλιο δεν παρίσταται ίσως ούτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε δεν μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σας. Είμαστε μεταξύ μας, μπορούμε απλώς να συζητήσουμε τις δικές μας θέσεις για το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Εγώ είμαι σκιώδη συγγήτρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, οπότε πολύ ευχαρίστω να σας παρουσιάσω τη δική μας θέση, τη θέση της ομάδας μου. Ε, χαιρόμαστε ε, για την πρότασή σας και συμφωνούμε με την αλλαγή της ονομασίας γιατί δεν νομίζω ότι η ονομασία αυτή ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του προγράμματος. Δηλαδή, ε, αλευθερία, δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα. Βέβαια, ίσως έτσι μακραίνει κάπως ο τίτλος, αλλά νομίζω ότι και τα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν μεγάλη σημασία στον ευρωπαϊκό χώρο ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. 0,7% είναι ε, του συνόλου του προπολογισμού πολύ μικρό προπολογισμό, παρόλο που η συνθήκη τη Λισαβόνα θεωρεί αυτό το τομέα όλο και πιο σημαντικό. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ομοφοβία, ε, μισαλλοδοξία κατά μειονοτήτων, Ρωμά, προβλήματα ελευθερίας έκφρασης στο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Είναι σημαντική εναρμόνιση των νομικών συστημάτων και ιδιαίτερη έμφαση στην δικαστική συνεργασία και στην ε, εκπαίδευση των αστυνομικών. Θα πρέπει να ε, παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινή μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου και να ανταποκριθούμε στις ε, ευνίδιες προκλήσεις όπως ήταν αυτή στη, της κρίσης στη Μεσόγειο. Προτείνουμε μία μικρή αύξηση του προϋπολογισμού, αμεληταία που παρόλα αυτά θεωρούμε ότι, ελπίζουμε τουλάχιστον, θα μπορέσει να καλύψει τα, πέναν, τα απαραίτητα βήματα. Περισσότερους πόρους χρειαζόμαστε, όπως είπατε κι εσείς, ε, για να αυξηθεί η ελαστικότητα. Επίσης η απλοποίηση είναι κάτι που έχουμε δεχτεί, η απλοποίηση στα διάφορα ε, ταμεία, κάτι που θα διευκολύνει τους ετούντες. Το συζητήσαμε και επ' του προγράμματος δικαιοσύνη και των δικαιωμάτων και ηθαγένεια. Θέλουμε κάποια συνέχεια αλλά και προβλεψιμότητα. Υπάρχουν διαφορετικοί στόχοι, έχουμε διαφορετικά δίκτυα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συμβάλλουν ιδιαιτέρως στους τομείς αυτούς και επιφέρουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Είναι σημαντικό όμως και για τους δικαιούχους να ξέρουν τι θα συμβεί μέσα σε αυτή την επιλογή, να υπάρχει μια προβλεψιμότητα λοιπόν δημιουργείται μια σταθερότητα. Έχουμε περισσότερα κονδύλια για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά για τα εξωτερικά σύνορα δεν έχει με αύξηση του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων ταμείων. Το πρόγραμμα δικαιώματα και Ιθαγένεια είπε ότι θα πρέπει να έχει απαραίτητη χρηματοδότηση για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων. Επίσης, όπως είπα, ο προϋπολογισμός του συγχωνευμένου προγράμματος Δικαιώματα και ηθαγένεια είναι μικρότερος από το άθροισμα των προϋπολογισμών των τριών προγραμμάτων που αντικατέστησε. Κρίμα. Βέβαια δεν έχουμε ακόμη σαφή ιδέα για το τελικό ποσό, αλλά αυτό το τμήμα της αύξησης που μας αναφέρατε στο συγκεκριμένο τίτλο ουσιαστικά σηματοδοτεί ε, μείωση του συνολικού ποσού. Επίσης, θα πρέπει τουλάχιστον ο συνολικός προϋπολογισμός να μην μειωθεί. Τα προγράμματα του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου πρέπει να είναι ε, συμπληρωματικά μεταξύ τους και να δώσουμε έφεση και στη συνέργεια. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία είναι η κατευθυντήρια γραμμή όλων αυτών των προγραμμάτων που θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Όπως είπαμε πολλές φορές σήμερα, υπάρχει πρόβλημα και με τους δείκτες. Είναι συνήθως ασθενείς οι δείκτες και οι στόχοι. Αν έχουμε περισσότερη ελαστικότητα, θα πρέπει τουλάχιστον να φροντίσουμε οι δείκτες να είναι σαφείς και ακριβείς για να μπορούμε πραγματικά να καταμετρήσουμε και να αξιολογήσουμε τις διάφορες δράσει και τα προγράμματα. Και οι στόχοι μας θα είναι συγκεκριμένοι. Αλλιώς δεν θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Σημαντικό θέμα είναι και τα ετήσια προγράμματα. Με την απλούστευση φοβούμαστε ότι θα μεληθούν κάποιοι στόχοι μέσα στην επταετία. Οι συμφωνούμε με την ελαστικότητα, είναι χρήσιμη. Και πάλι προτιμούμε ε, τα, τις κατεξουδότηση πράξης για το πρόγραμμα ε, ισότητας και δικαιώματα και ηθαγένεια. Αυτά είναι λοιπόν κάποια προκατακτικά σχόλια. Πιστεύω ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία και στο μέλλον. Κρίμα που δεν είναι παρόντες εδώ εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ελπίζουμε τουλάχιστον στην επόμενη συζήτηση κάποιος να παρουσιαστεί. Κύριε Μπρόζ, έχετε το λόγο. Κυρία Χολμάγερ. Ε, η κυρία Χολμάγερ περίμενε σχόλια από του συναδέλφου. Ε, γύρισε και κοίταξε λοιπόν και έμεινε ευρώντη γιατί μόνο εγώ είμαι εδώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Φαίνεται ότι η, ε, δαπάνη σημαντικών ποσών των φορολογουμένων δεν είναι αρκετό λόγο για να κρατήσει του συναδέλφου μέσα στην αίθουσα. Λοιπόν, θα μιλήσω ξεκάθαρα γιατί στην προηγούμενη συνεδρίαση με ευχαριστήσατε, κυρία Πρόεδρε, γιατί ε, επέκτηνα τα, την προσθήκη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και σε ε, υπηκό χωρών. <laughs> Δεν ήταν δική μου πρόταση. Εγώ το, την αποδοκίμασα. Απλώ ανέφερα δικό σα εδάφιο από την δική σας έκθεση. Επίσης, ό,τι αφορά την παράγραφο 4, περιλαμβάνει μνήμα στην επανεγκατάσταση ε, και στα μέτρα επαναπατρισμού ή επιστροφής και μάλιστα στην ίδια παράγραφο. Ερωτώ λοιπόν πόσα κονδύλια θα δοθούν για μέτρα επιστροφής σε σχέση με την επανεγκατάσταση. Ε, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και πολλά αυτά τα χρήματα με βάση τις μαρτυρίες του εκτελεστικού διευθυντή της Frontex που παρακολουθήσαμε πριν από τρεις εβδομάδες γιατί οι λαθρομετανάστες ε, ανακαλύπτονται και συλλαμβάνονται από την Frontex, αλλά δεν κρατούνται. Του δίνουν ένα χαρτί που λένε ότι σε τόσε μέρε πρέπει να εγκαταλείψουν το έδαφο, αλλά δεν του παρακολουθούν, ούτε ε, γίνεται κάποιο έλεγχο, ή δεν υπάρχει υποχρεωτική επιστροφή. Και φαντάζομαι κανένα δυο από αυτού <laughs> δεν πολύ παίρνουν στα σοβαρά αυτό το χαρτί. Εκτό κι αν εγώ είμαι πια δύσπιστο και καχύποπτο. Σα ευχαριστώ κύριε Μπρόνς. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει το λόγο αλλά δεν υπάρχουν και πολλοί με στην αίθουσα. Κυρία Χολμάγερ, δεν ξέρω αν έχετε σχόλια μετά από αυτά που ακούσατε. Τι να σας πω, συμπερασματικά να σας πω ότι πραγματικά για τις τροπολογίες, για την κατάθεση τροπολογιών θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τις προτάσεις μας, όπως είπε και ο κύριος Μπρόγκ στο άρθρο 4 προσπάθησα να συνοψίσω όλα αυτά, γιατί καταλαβαίνετε ότι στα πλαίσια μίας γνωμοδότησης, όταν έχουμε δηλαδή λιγότερο από μία σελίδα, τρία τέταρτα της σελίδας στη διάθεσή μας, δεν μπορούμε να μπούμε σε περισσότερη αιτιολόγηση και περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν προλαβαίνω δηλαδή ε, να εξηγήσω περισσότερο, δεν έχω το χώρο και τη δυνατότητα. Δεν ε, μου λείπει η επιθυμία, αν θέλετε, αλλά έχω τρία τέταρτα μία σελίδα στη διάθεσή μου. Τι μπορώ να πω παραπάνω για όλες αυτές τις κατηγορίες. Σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία σε όλα αυτά τα συνοδευτικά μέτρα. Σίγουρα θα πρέπει να βοηθήσουμε τις ε, πατρίδες, ε, τα χωριά αυτών των ανθρώπων όταν επαναπατρίζονται για να μπορέσουν να μείνουν εκεί. Αυτό που πραγματικά θα έλεγα εγώ στα γερμανικά, αλλά είναι κάτι που βεβαίως δεν μπορώ να το μεταφράσω εύκολα, είναι ότι προσπάθησα να κάνω μια επιλογή η οποία δεν είναι εύκολο να γίνει. Βεβαίως, αν εσείς μπορείτε να γυρίσετε σπίτι σας και να έχετε μια καλύτερη ζωή, θα το κάνετε. Αλλιώς δεν νομίζω ότι αυτό είναι μια ευνοϊκή προοπτική. Πάντως χαίρομαι γιατί μπορέσαμε να έχουμε μια πολύ ε, επικοδομητική συνεργασία και συζητήθηκαν όλες, ακόμα και πιο ακραίες ε, προτάσεις. Ευχαριστώ κυρία Χολμάιερ. Δεν βλέπω κάποιον εδώ παρόντα στην αίθουσα να θέλει να πάρει το λόγο. Τι να κάνουμε άλλο από το να καθορίσουμε την ε, ημερομηνία υποβολής των τροπολογιών, Τετάρτη 11 Ιουλίου το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στις 3 Σεπτεμβρίου. Μάλλον θα εξετάσουμε, συγγνώμη, και 19 και 20 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή. 19 και 20 Σεπτεμβρίου η ψηφοφορία στην Επιτροπή. Περνάμε στο επόμενο σημείο που επίσης θα μας παρουσιάσει η κυρία Χολμάιερ. Είναι το σημείο 15 που αφορά επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών και κατάργηση της απόφασης πλαίσιο 2005 κάθετος 222. Πρόκειται για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Υπάρχει εδώ ήδη μια διαδικασία τριμερούς διαλόγου. Κυρία Χολμάιερ, με ακούσατε? Η συγγήτρια θα μας ενημερώσει για το τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων σε αυτόν τον τίμερη διάλογο. Στις 4 του μηνός έλαβε χώρα. Σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης εβδομάδας, απόφαση της συνδιάρκειας των Πρόεδρων, έχει διακοπεί η διαπραγμάτευση και η συζήτηση με το Συμβούλιο για θέματα που αφορούν το πακέτο Σέγγεν. Κυρία Χολμάιρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως προς το περιεχόμενο αυτής της οδηγίας, πρώτης οδηγίας, πρόκειται ουσιαστικά για σοβαρές επιθέσεις και εγκλήματα στα συστήματα πληροφοριών να υπάρξει μια σύγκληση των συστημάτων και των προβλέψεων και όσον αφορά τις κυρώσεις αλλά και να υπάρξει μια σύγκληση των διαφόρων συστημάτων. Σήμερα δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει κανείς, ε, όπως ξέρετε, τα σύγχρονα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Η τεχνολογία εξελίσσεται καθημερινά και με ραγδαίους ρυθμούς. και αυτό και προσπαθήσαμε να διαλέξουμε μια ουδέτερη διατύπωση έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι διάφορες τεχνολογίες και την ίδια ώρα να μπορέσουν να καλυφθούν όλες οι εγκληματικές πράξεις άσχετα με το πώς και πότε έχουν ε, εξελιχθεί διάφορες τεχνολογίες. Τέλος Μαρτίου του 2012 ψηφίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία. Υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις, αν θέλετε, τρεις άξονες. Πρώτον, δεν θέλουμε να υπάρξει υπερβολική χρήση του χαρακτηρισμού ποινικό αδίκημα ή έγκλημα. Δεν θέλουμε δηλαδή να συμπεριληφθούν και πολύ μικρές οι ελάσσονο σημασία πράξεις, οι ελάσσονος σημασίας πράξεις, ε, αδικήματα, θέλουμε να συμπεριληφθούν σε μία άλλη κατηγορία, να μην δηλαδή υπόκεινται σε ποινή. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ μας άκουσε το Συμβούλιο. Το θέμα της πρόληψης όμως που προϋποθέτει καλύτερη συνεργασία, καλύτερη παρακολούθηση της επιβολής των ποινών και σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών φορέων και των ευρωπαϊκών υπηρεσιών και οργανισμών. Εδώ θα πρέπει να ληφθούν πολύ συγκεκριμένα μέτρα στα πλαίσια της προληπτικής πολιτικής, δηλαδή κάποια ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας για όλα τα συστήματα, καθότι για να χαρακτηριστεί ως αξιόπινο ένα δίκημα και να φτάσουμε στην πραγματική κύρωση θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις προηγούμενες ε, φάσεις της διαδικασίας. Αυτή λοιπόν είναι η στρατηγική μας και αυτό είναι και ο σκοπός αυτής της οδηγίας και ενδεχομένως ενός κανονισμού. Η Επιτροπή παρόλα αυτά αντίδρα με σχετική βραδύτητα όσον αφορά το ντρεμερή διάλογο. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Προεδρία της Δανίας. Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου τέτοια προσπάθεια να καταλάβει και να πλησιάσει τις θέσεις μας. Πραγματικά οι συναντήσεις που είχαμε με την Δανική Προεδρία στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου ήταν εξαιρετικά επικοδομητικές. Προσπάθησαν πραγματικά να καταλάβουν αυτά τα οποία λέμε και αυτά τα οποία ε, τους προτείνουμε. Ευχαριστώ και την Προεδρία της Πολωνίας και της Ουγγαρίας για την προετοιμασία που ε, έκαναν για αυτήν την ε, υπόθεση. Είχαμε πολύ καλή ανταλλαγή επίσης και με την Επιτροπή όσον αφορά το περιεχόμενο τουλάχιστον. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό και καταφέραμε τελικά στην τελευταία συνάντηση που είχαμε να περάσουμε πολλές από τις θέσεις του Κοινοβουλίου και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και με μεγάλη πλειοψηφία μπορέσαμε να πετύχουμε κοινέ θέσεις στα περισσότερα από αυτά που προτείναμε. Ήθελα επίσης να σας πω ότι όσον αφορά το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής συμφωνίας, Όσον αφορά το περιεχόμενο, μπορέσαμε πραγματικά να περάσουμε κάποιε από τι θέσει μα, όπως τον καλύτερο ορισμό, τη διασαφήνιση ποιών δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε ποινικέ διώξει και κυρώσει. Οι ορισμοί, αν θέλετε, minor cases, ελάσσονο σημασία υποθέσει. επίσης νέοι οι οποίοι καλή την πίστη αν θέλετε διαπράττουν κάποιο ε, κάποια παράβαση έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη πρόληψη, καλύτερη ενημέρωση κτλ. και να υπάρχει διάκριση μεταξύ αυτών των υποθέσεων και των αξιόπινων. Συνεργασία με την Ινίσα, την Europol, την Eurojust υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σε εθνικό επίπεδο επαφές. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί αν αποφασίσουμε να υπάρχει ένα μεγάλο κέντρο για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν σημεία αναφοράς παντού σε όλες τις χώρες μέλη. Επίσης, ειδικά συστήματα όσον αφορά τη σαφή παρουσίαση των ευθυνών, συστήματα ασφάλειας, το θέμα της ε, ταυτοποίησης του αυτούργου σε περίπτωση που αυτός έχει χρησιμοποιήσει μια άλλη ταυτότητα από την πραγματική του για να διαπράξει ένα αξιόπινο, ε, μια αξιόπινη πράξη. Το θέμα λοιπόν της ευθύνης και της ασφάλειας και πραγματικά θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε όλα αυτά τα σημεία σε καλή ε, οδό. Οι δικές μας επιθυμίες πραγματικά έχουν ληφθεί υπόψη. Το θέμα είναι αν το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίξει αυτά που έχει ζητήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό δεν είναι θέμα μου στο Συμβουλίο, είναι δικό μας θέμα. Κατά κάποιο τρόπο έχουν έρθει τα πράγματα πάνω κάτω. Ζητούμε κάποια πράγματα, το Συμβούλιο τα δέχεται και μετά εμείς δεν τα υποστηρίζουμε. Εν πάση περιπτώσει, ε, ευχαριστώ πολύ το Συμβούλιο γιατί δεν μας εκδικείται, δεν χρησιμοποιεί αυτή την αδυναμία μας και πιστεύω ότι σε μεγάλη πλειοψηφία, επαναλαμβάνω, οι προτάσεις που κάναμε και έγιναν δεκτές θα υποστηριχτούν μέχρι το τέλος. Εγώ πραγματικά ευχαριστώ γιατί η Προεδρία της Δανίας έκανε εξαιρετική εργασία στο αυτό. Σας ευχαριστούμε κυρία Χολμάγερ για την έκθεσή σας και την ενημέρωση. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Θεανικής Προεδρίας. Γιατί εγκομιάσατε την Προεδρία για την συνεργασία και τις προσπάθειές της για το θέμα αυτό. Το τονίσατε κυρία Χολμάιερ. Οπότε Φαντάζομαι ότι κάτι θα θέλει να πει εκπρόσωπο τη Ελληνική προεδρία και ίσως ε, να ακούσουμε και κάποιον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Προεδρία. Στο πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρου του Συμβουλίου είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να σα καταθέσω ότι χθε στο Κοροπέρ εξετάσαμε αυτό το θέμα και υπήρξε έγκριση του, κίνημα, του κειμένου όπως έχει αυτή τη στιγμή και συμφωνήσαμε σε αυτό το κείμενο Συνεπώς, ευτυχώς πρόεδρε, θα δείτε μια επιστολή η οποία θα έρθει από το κοροπέρι, η οποία, η επιστολή αυτή, θα εγκρίνει το κείμενο που έχουμε αυτή τη στιγμή αναχείραση. Κάτι άλλο τώρα. Υποστηρίζω τον εισηγητή, ο οποίος έχει πει ότι βρήκαμε μια σωστή συμβαστική λύση και πιστεύω πως με αυτό, μεταξύ αυτού του τριλόγου θα έλεγα, τριπλού διαλόγου, νομίζω πως καταλήξαμε και χάρη στις προσπάθειες του Κοινοβουλίου γίναμε κατέστημεν ικανοί να εισάγουμε πολλά πράγματα που έχει προβάλλει το Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν, ε, έτσι πρέπει να είναι οι διαπραγματεύσει και οφείλω να ομολογήσω πως Είμαι ευγνώμων στην εισηγήτρια και την ομάδα της που μπόρεσε να δημιουργήσει τόσο καλή ατμόσφαιρα για αυτές τις διαπραγματεύσεις μία με μία πολύ επικοδομητική προσέγγιση. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιό που υποστήριξε αυτό το τρίλογο θα έλεγα. Έτσι. Ευχαριστίες και πάλι στους μεν και στους δε βεβαίως αυτό Ξέρετε, είναι νεκρεμότητα αυτό το θέμα, μας αφήνει με αυτή τη γεύση στο σώμα. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι αυτό το θέμα που εκκρεμεί φαχύτερο δυνατόν θα επιληθεί, ούτως ώστε όλος αυτός ο φάκελος και η υπόθεση αυτή να περιοθεί τελειωτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έχει να μας πει η Κομισιόν παρακαλώ, θα θέλατε και εσείς να πείτε. Πολύ σύντομα πρόεδρε για να πω το εξή. Η Κομισιό χαίρεται πάρα πολύ γι' αυτό το επιτυχές αποτέλεσμα μεταξύ αυτού του τριπλού διαλόγου που έχει γίνει. Αυτό είναι ένα καλό αποτέλεσμα, όπως είπα, και το υποστηρίζουμε. Ακόμη, θα έλεγα, είναι, είναι ένα μέρος για τα JICS και θα επανέλθουμε με περαιτέρω προτάσεις στο μέλλον για δραστηριοποίηση και διότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν όσον αφορά το ποινικό δίκαιο καθώς επίση και το κυβερνοχώρο χαιρόμαστε με τα επιτευχθέντα μέχρι τούτου μέχρι τούδε. και βεβαίως ό,τι άπτεται με το Σέγγεν προφανώς είναι θέματα τα οποία έχουν σχέση με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο. Η Κομισιόν λοιπόν προσβλέπει το γενικότερο αυτό το θέμα θα, ότι θα πρέπει να επιληθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μεταξύ αυτών των των δυο δύο οργάνων. Ευχαριστώ. Υπάρχουν δύο-τρία μέλη οι οποία θέλουν να μιλήσουν. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ο κύριος Σένσιο έχει το λόγο παρακαλώ πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τη Μόνικα Χολμάιερ και να ενημερώσω την Επιτροπή μας ότι είναι πραγματικά μια καταπληκτική αγωνίστρια η Μόνικα και μπορούμε να στηριχθούμε πάνω της και να είμαστε βέβαιοι ότι όταν αναλαμβάνει ένα τόσο σημαντικό θέμα θα το φέρει σε αίσιο Ήταν καρποφόρα η συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια του τριμέρους διαλόγου. Βέβαια, την περισσότερη δουλειά την έκανε η συγγήτρια, που πραγματικά κατάφερε να λάβει υπόψη τα αιτήματα όλων των πολιτικών ομάδων στην τελική της έκθεση. Χαίρομαι που μετά από τους τρεις τριμερείς διαλόγους ε, καταλήξαμε σε συμφωνία και με το Συμβούλιο και πιστεύω ότι η συμβαστική λύση του τελευταίου τριμερούς διαλόγου είναι ικανοποιητική. Γιατί λαμβάνονται υπόψη τα βασικά μας αιτήματα, όπως η εφαρμογή σε οργανισμούς και υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που σχετίζονται ε, με την πάταξη του εγκλήματος, όπως είναι η Europol και η Eurojust. Προσδιορίζεται ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα προκειμένου να αποτραπούν τέτοιες επιθέσεις σε συστήματα πληροφόρησης. Είναι απαραίτητος και ο συντονισμός σε διεθνές επίπεδο, αλλιώς είναι αδύνατο να καταπολεμηθεί η κυβερνοεγκληματικότητα. Ένα άλλο θέμα ιδιαίτερα προσφυλές που δέχτηκε το Συμβούλιο είναι η βελτίωση του πλαισίου θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια της καταπολέμησης της ε, κυβερνοεγκληματικότητας. Επίσης, ε, τα κράτη-μέλη και οι εθνικές αρχές ε, οφείλουν και αυτές να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, χαίρομαι που ε, γίνεται διαφοροποίηση των κυρώσεων και είναι πιο αυστηρές ανάλογα με τις παραβάσεις, όπως και οι αποζημιώσεις. Οι επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές που δημιουργούν πολύ σοβαρές ζημιές θα ε, τιμωρούνται με φυλάξη τουλάχιστον 5 ετών. Βέβαια, κάποιες ε, προτάσεις μας δεν έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο, όπως ε, την ευθύνη των νομικών προσώπων να προστατεύσουν τα συστήματα πληροφορικής της. Αυτό περιλήφθηκε μόνο στο προήμιο της οδηγίας, με μια πολύ πιο αδύναμη διατύπωση από αυτή που ζητούσαμε εμείς. Επίσης, το θέμα της ε, ενημέρωσης ε, για θέματα κυβερνοκληματικότητας δεν είναι αρκετά εμφανές στην οδηγία, αλλά ελπίζω να αποτελέσει το αντικείμενο ξεχωριστό της ε, πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγένει το κείμενο είναι ικανοποιητικό και πιστεύω ότι η νέα οδηγία πραγματικά θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε τις διάφορες μορφές επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφορικής. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Δανική Προεδρία για την προσέγγιση που υιοθέτησε και τη συνεργασία που είχε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ευχαριστώ και θα σα ευχαριστήσω την προλαλήσατε καθώς επίσης και τη Μόνικα για την εργασία που επιτέλεσε και που είναι μακρόπνοη εργασία και μας πήρε σε μια πολύ καλή συμβιβαστική λύση συγχαρητήρια και χαιρόμαστε όλοι. Και είναι περισσότερο και πολύ και ευχάριστο το κείμενο αυτό αυτό. Θα ήθελα ακόμη να σχολιάσω πως πραγματικά υπάρχει ένα μπλοκαριστή ακόμη το κείμενό τη από, τον προ, από τους Προέδρους. Εσείς δεν φταίτε κύριε Πρόεδρε, σαν δικό μας Πρόεδρος, αλλά θα ήθελα να σας πω πως υπάρχει ένα ντοσιέ το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή και το οποίο θα πρέπει να έρθει στην Ολομέλη και το Προεδρείο, το Σύνος των Προέδρων είχε απάντησε πως ότι μπλοκάρεται και νομίζω ότι αυτό το, το μπλοκάρισμα δεν είναι η καλύτερη απάντηση η οποία θα πρέπει να δοθεί σε αυτό το θέμα και θα πρέπει να το ξέρει και η Δανική Προεδρία και το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να το φέρει προ συζήτηση. Και δημοσιονομική και οικονομική. Ε, πράγμα το οποίο θα είχε πολύ χειρότερα αποτελέσματα για το Συμβούλιο από ότι αυτό. Η κυβερνό εγκληματικότητα είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Υπάρχει μια επιτροπή ε, ΚΡΙ, η οποία είναι ειδική για την έρευνα του θέματος αυτού για την κυβερνό εγκληματικότητα και άπτεται όλων των πολιτών και θα πρέπει να δούμε πραγματικά πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντιδράσει πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω πως είναι η καλύτερη υπόθεση που θα μπορούσαμε να κάνουμε για ένα τέτοιο κείμενο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή αναχέδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μπρόγκς παρακαλώ, έχει το λόγο. Really... αυτό. Uh, ε, ένα θέμα προς το υπόβαθρο της πρότασης αυτής παρά ως προς την ουσία. Έχουμε ιδιώτες ή ομάδες που επιτίθενται σε συστήματα πληροφορικής, αξιολύπητη αυτή η δράση και φυσικά θα πρέπει να αναλυφθούν δράσεις από τις αρχές. Εμένα με ε, ανησυχεί κάπως η αντίδραση των κυβερνήσεων σε ό,τι αφορά τα συστήματα πληροφορικής άλλων κυβερνήσεων. Και δεν είναι απλό σενάριο η Γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ και η ΙΠΑ ε, επιτέθηκαν στο, στο πρόγραμμα πληροφορικής ε, του πυρηνικού συστήματος του Ιράν. Και μπορεί να λένε μερικοί ότι είναι δικαιολογημένο. Δικαιολογημένο, ξεδικαιολογημένο είναι γεγονός. Και η Κίνα μπλοκάρει κάποιε ιστοσελίδε, παρόλο που δεν επιτίθεται σε συστήματα πληροφορικής άλλων κυβερνήσεων. Η Κυρία Χολμάγερ, από την έρευνα που έκανα προετοιμάζοντα την έκθεση γνωρίζει αν κάποιε ευρωπαϊκές χώρες ή η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση επιτίθεται συστήματα πληροφορικής τρίτων χωρών ή μήπω ε, αν ε, υπάρχει δράση τρίτων χωρών κατά συστημάτων πληροφορικής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωση. Δεν αναφέρομαι φυσικά σε πλήρω δικαιολογημένη δράση κατά απαταιώνων ή όσων διακινούν παιδική πορνογραφία ή άλλων εγκληματιών, γιατί είναι <laughs> αυτονόητο ότι δικαιολογούνται επιθέσει και μπλοκαρίσματα τέτοιων ιστοσελίδων. Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τις, να προσθέσω τις ευχαριστήσεις μου στον κύριο Χολμάγερ για την εργασία την οποία έχει επιτελέσει η εγκληματικότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό αναφέρθηκε. Είναι κάτι το οποίο ε, θα εξεταστεί από την Επιτροπή ΚΡΙΜ, η οποία είναι ειδική επί του θέματο αυτού. Ωστόσο, θα σχολιάσω λέγοντα το εξή, ότι η δραστηριότητα που ανέλαβε το Κοινοβούλιο μα ε, και το Σύμβουλο των Προέδρων ε, η ομάδα μου αντιτάχθηκε τη δραστηριότητα που ανέλαβε, όπου η συνδιάσκεψη των Προέδρων έχει αναλάβει διότι διότι παίρνει πραγματικά μερικά θέματα και αποφεύγει τη δυνατότητα που μπορούμε να έχουμε σε συνεργασία με το Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι πεδαριώδες αυτό το οποίο έχει γίνει. Και ακόμη κάτι, ότι θα εμφανιστεί εν τελική αναλύση στο Κοινοβούλιο ηλίθιο ενώπιον των τρίτων και η νομική άποψη η οποία θα δοθεί από το κείμενο, από το νομικό προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο δρά μέσα στα δικά της δυνατότητες που έχει και δεν μπορεί να αποσύρουμε αυτή τη δυνατό ε, να αποσύρουμε εμείς αυτή τη δυνατότητα συνεργασία που έχουμε. Αυτό με εκπλήσει πάρα πολύ και αυτό, αν καταπέσει τελικά, θα είναι πραγματικά ντροπή, θα είναι κρίμα και θα είναι πάρα πολύ καταστροφικό θα ήθελα απλώ να καταγραφεί αυτό το οποίο σας έχω πει και να μπει στα πρακτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σάνρεχτ, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη γιατί καθυστέρησα. Συνήθως καθυστερούμε στην ημερησία διάταξη, γι' αυτό ήρθα και λίγο καθυστερημένος. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά έχω λίγο χρόνο από ό,τι φαίνεται για να πω δύο λόγια. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η συνεργασία είναι πάντα επικοδομητική με την εισηγήτρια, πάντα δίνει την εντύπωση τουλάχιστον ότι ακούει, ότι λαμβάνει υπόψη της αυτά που ακούγονται. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, βέβαια τα πράγματα δεν είναι άσπρο-μαύρο. Το θέμα είναι ότι από τη μία μεριά έχουμε την οδηγία για τις ποινικέ κυρώσεις κατά των εγκληματικών πράξεων και από την άλλη μεριά ο νομοθέτης πρέπει σαφώς να πάρει κάποια μέτρα όσον αφορά τη διασφάλιση της ασφάλειας και να δώσει και κάποια κίνητρα έτσι ώστε να οδηγήσει σε περισσότερη ευαισθητοποίηση και ανάληψη ευθυνών από όλους αυτούς οι οποίοι πολλές φορές ε, είτε κάνουν σφάλματα είτε πέφτουν στις παγίδες των κενών ε, της ε, έλλειψης κάθε νομοθεσίας παραδείγματο χάρη. Αυτό εμείς σαν πράσινοι θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και όσον αφορά τη λεγόμενη white hat hacking, δηλαδή αυτές τις πράξεις οι οποίες γίνονται καλή την πίστη. Κάποιοι δηλαδή μπαίνουν σε κάποια συστήματα πληροφοριών χωρίς παρόλα αυτά να έχουν την πρόθεση να διαπράξουν ένα αξιόπνο, μια αξιόπνη πράξη. Παρόλα αυτά, ε, συνειδητά ή ασυνείδητα κάνουν κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να το χαρακτηρίσουμε διαφορετικά. Εν πάση να ξεκινήσουμε μια συζήτηση γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε παρόλα αυτά δυσκολίες να δεχτούμε το αποτέλεσμα των ε, διαφόρων και χαρήκαμε ιδιαίτερα όταν είδαμε ότι θα περάσουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Δεν ξέρω βέβαια τι δυνατότητες έχουμε τώρα με αυτό που αποφασίστηκε γενικότερα για το πακέτο Σέγγεν να συνεχίσουμε συζητήσεις για το θέμα αυτό. Τι περιθώρια λιγμό έχουμε. Εμείς ε, πολύ θα θέλαμε να δούμε αν υπάρχουν δυνατότητες εξέλιξης ή αν θα παραμείνουμε στην παρούσα κατάσταση. Ευχαριστώ πάντω πάρα πολύ για την συνεργασία που είχαμε. Πρόεδρος, ωραία, εισηγήτρια. Να ακούσουμε τα τελικά σας σχόλια. Ακούσατε τους μεν και τους δε, μπορείτε να απαντήσετε. Ναι, καταρχήν να απαντήσω σε δυο τρει ερωτήσεις. Κύριε Μπρόγκ, όσον αφορά τις επιθέσεις κρατών κατά συστημάτων. Κοιτάξτε, ο Τίμωθη Κέρκελ έχει δώσει ένα συγκεκριμένο νομικό έγγραφο γι' αυτό. Δεν μπορούμε εμείς να ασχοληθούμε με το θέμα επιθέσεων κρατών κατά άλλων κρατών. Το συζητήσαμε, ακολούθησε μάλιστα μια έντονη αντιπαράθεση. Ε, αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι στην οδηγία αυτή για τα ποινικά δίκαια δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν αυτές οι περιπτώσεις και σαφώς εμείς εκφράσαμε την επιθυμία μας να ε, ρυθμίσει το θέμα αυτό των επιθέσεων κρατών καρακρατών το διεθνές δίκαιο. Αυτή είναι η λογική, αν θέλετε, η οποία επικράτησε. Το τι κάνει τώρα η Κίνα, τι κάνει η Ρωσία, ολόκληρη σειρά επιθέσεις έχουν ε, γίνει. Αν αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά, καταλαβαίνετε ότι η εργασία που θα πρέπει να επιτελέσουμε θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Εν πάση περιπτώσει, εδώ πρόκειται για ένα άλλο θέμα. Δεύτερον, κύριε Άλμπρεχτ, και εμείς δεν είμαστε ευτυχείς γιατί αυτή η οδηγία είναι αυτή τη στιγμή αυτή που πλήττεται, καθώς και όλες οι άλλες πρωτοβουλίες ε, που ακολουθούν. Όλα αυτά σταμάτησαν τώρα. Υπάρχουν και θέματα ελάχιστων προτύπων, υπάρχουν και τα θέματα των κινήτρων για τους νέους, ε, τους λεγόμενους white hat hackers σαφώς και εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι το θετικό, όχι μόνο περιορισμούς και προειδοποίηση. Το είπα στα εισαγωγικά μου σχόλια, λέγοντας ότι εκφράζω την απογοήτευσή μου γιατί όλα αυτά ακόμα δεν συμπεριλαμβάνονται. Αλλά βεβαίως το κείμενο ήταν πολύ σύντομο. Το θέμα του ποινικού δικαίου στην Ευρώπη και το εάν και πόσο μπορούμε να συγκλίνουμε είναι γνωστό. Βεβαίως, η περίπτωση των περιπτώσεων ε, ελάσσονος σημασίας αναφέρεται, αλλά όχι βεβαίως στο κυρίως κείμενο. Αυτές οι περιπτώσεις ε, ελάσσονος σημασίας είναι περιπτώσεις τις οποίες βεβαίως αναφερόμαστε, αλλά Πρόκειται για περιπτώσεις όπως παραδείγματο χάρη κάποιος ο οποίος μπορεί να προσχωρήσει και να παραβιάσει ένα σύστημα, αλλά η... τα πλήγματα τα οποία επιφέρει δεν είναι τόσο σημαντικά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις αναφερόμαστε, όχι μόνο της μη εθελοντικής παραβίασης. Θέλουμε λοιπόν να ενσωματώσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις χωρίς βεβαίως να μπορούμε να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Θέλουμε να δημιουργηθούν παραδείγματος χάρη προγράμματα τα οποία θα συμπεριλάβουν και όλους αυτούς τους νέους ε, hackers ε, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους στον τομέα της πληροφορικής για να δοκιμάσουν τα προγράμματα. Τα νέα προγράμματα δηλαδή κατά κάποιο τρόπο δοκιμάζονται από τους νέους hackers για να δούμε κατά πόσο είναι απαραβίαστα. Αν λοιπόν εμείς δημιουργήσουμε αυτά τα προγράμματα και τους καλέσουμε, κατά κάποιο τρόπο προλαμβάνουμε τον κίνδυνο παραβίασης εκούσιας ή ακούσιας Θέλουμε λοιπόν να έρθουμε σε επαφή με αυτές τις κατηγορίες νέων ανθρώπων, σε αυτές τις κατηγορίες που μέχρι τώρα δεν είχαμε επαφές. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, άκουσα την άποψη του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο θέλει να συμπεριληφθούν αυτές οι περιπτώσεις ελάσσονος σημασίας, όπως τις ονομάζουν, και περίπου δυόμιση ώρες πρέπει να σας πω μιλήσαμε για αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Δυόμιση ώρες για μια αιτιολογική σκέψη. Εν πάση περιπτώσει βρέθηκε μια διατύπωση και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί οι συνάδελφοι από τους πράσινους θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτοί σε αυτή τη διατύπωση έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ένα ενιαίο μήνυμα προς τα έξω. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους, ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν και βεβαίως υπήρχαν και περίπλοκα θέματα. Ευχαριστώ όλους τον Άλβαρο, Άλμπρεχτ και όλους όσους συμμετείχαν σε αυτήν την ε, πολύ έντονη συνεργασία που είχαμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως τελειώσαμε πραγματικά αυτή τη συζήτηση. Είναι ένα σχέδιο. Θα υπάρχει ένα, ένα briefing όσον αφορά τον τρίλογο, μια ενημέρωση και νομίζω πως πραγματικά είναι αρκετά για, προς το παρόν και προσδοκούμε να υπάρξει και περαιτέρω εξέλιξη και τα θέματα τα οποία το αφορούν το Eurojazz με του νέου εκλεγμένου, του, προ, του νέου εκλεγέντος ε, της κυρίας Κόνη να εκλεγήσεις. Δεν είναι ακόμη εδώ. Σε 11.30 θα ξεκινήσει. Υπάρχει λοιπόν μια διακοπή που θα κάνουμε για 5 λεπτά. Θα ξεκινήσω σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.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

Σταματήστε παρακαλώ. May have your attention, please. Και λίγη προσοχή. We have one hour to go. Μία ώρα μας έχει μείνει ακόμη. We're to make good use of it. Και θα την αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική καλεσμένη σήμερα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, την οποία και καλωσορίζουμε θερμότατα. Πρόκειται για την κυρία Μισελ Κόνιγκς, την εκλεγήσα πρόεδρο της Eurojust. Constellation. Είναι μία από, τους οργα... μία από τις υπηρεσίες ε, του αστερισμού της πολιτικής ε, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Τον προηγούμενο πρόεδρο τον είχαμε πολύ συχνά σε ακράσεις. Η κυρία Μισελ Κόνιγκς μόλις ανέλαβε τα καθηκόντά της. Της ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, καθήκοντα Προέδρου της Eurojust. Θα μας παρουσιάσει τώρα την ετήσια έκθεση της Eurojust. Η έκθεση αυτή επισημαίνει τις δραστηριότητες της Eurojust, αυτής της πολύ σημαντικής υπηρεσίας, του πολύ σημαντικού οργανισμού που ε, έχει 10 χρόνια ζωής και όλο και αυξανόμενη σημασία. Ο αριθμός των υποθέσεων που απασχόλησαν την Eurojust ε, το 2011 ήταν 1441 και γίνονται και πολλές συντονιστικές ε, συναντήσεις. Από το 2010 στο 2011 διπλασιάστηκαν από 120 200 και οι τέτοιες συντονιστικές συνεδριάσεις. Μάλιστα η Eurojust ε, συμμετέχει σε ερευνητικές ε, ομάδες των κρατών μελών προβλέπει και χρηματοδότηση για τέτοιου είδους διερευνητικές ε, ομάδες. Και πριν από λίγο στο Λουξεμβούργο έλαβε χώρα ένα πολύ σημαντικό σεμινάριο με θέμα την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Ασφάλειας Δικαιοσύνης και ελευθερία στα πλαίσια ποινικού δικαίου για αστυνομικέ και δικαστικέ έρευνε ε, και συνεργασία κυρίω αστυνομική και δικαστική συνεργασία γιατί είναι σημαντικό να προσάγονται στη δικαιοσύνη διασυνοριακά εγκλήματα, αυτούργοι διασυνοριακών εγκλημάτων, όπως προβλέπει το ε, σχετικό άρθρο της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το θέμα ε, πλέον υπόκειται στις νομοθετικές αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άρα της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών της δικής μας. Το θέμα της λειτουργία τη της Eurojust το κρίνουμε μέσω της ετήσια έκθεση που υποβάλλει κάθε χρόνο η υπηρεσία αυτή. Θα γίνει μια αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των επιχειρησιακών της δράσεων, τη διοικητική της οργάνωση, έκβαση της μελέτης που έγινε για τη Eurojust από την Deloitte πώς θα εφαρμοστεί και σίγουρα η Eurojust θα μπορούσε να έχει πολύ πιο στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τη δική μας Επιτροπή δίνοντας κάποιες συμβουλές για προτινόμενα νομοθετικά μέσα, όπως είναι η διγεία για το πάγωμα και την κατάσχεση, η δίμευση το, των κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Κόνιγκς, μόλις χθες στη συνεδρίαση των συντονιστών βασίσαμε να στείλουμε αποστολή της Επιτροπής μας στην έδρα της Eurojust, το επόμενο φθινόπωρο, στη Χάγη. Και φυσικά θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον όλες τις εξελίξεις της Eurojust προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 86 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Όχι μόνο για να εξασφαλιστεί η προστασία των οικονομικών συμφερόντων και δημοσιονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για να αντιμετωπιστούν περισσότερο και πιο αποτελεσματικά τα διασυνοριακά εγκλήματα. Αυτές είναι οι αναμενόμενες εξελίξεις στο έργο της Eurojust που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Και σίγουρα όσοι λάβουν το λόγο θα αναφερθούν σε όλα αυτά τα θέματα, αλλά και σε πολλά άλλα στη συζήτηση που θα ακολουθήσει τις παρουσίασεις. Κύριε Κόνιγκς, έχετε το λόγο. Καταρχήν σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε και σας ορίζουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά για τα πολύ ευγενικά εισαγωγικά σας σχόλια. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που έρχομαι στην Επιτροπή σας για να δώσω μια γενική επισκόπηση της ετήσιας μας έκθεσης για το 2011. Ε, έχουμε μοιράσει περίπου 100 ε, αντίγραφα αυτής της έκθεσης στην Επιτροπή, αλλά υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή πρόσθετη έκθεση σε 13 γλώσσες, με στόχο να μεταφραστεί και στις 23 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε αποφασίσει εδώ και καιρό να επικεντρωθούμε στις επιχειρησιακές δραστηριότητες της Eurojust και αυτές κυρίως να περιγράψουμε στην έκθεση. Και επίσης αποφασίσαμε να υπογραμμίσουμε την προστιθέμενη αξία της Eurojust, ιδιαίτερα στον τομέα της καταπολέμησης του διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος όπως είπατε κι εσείς, έχουν φτάσει στην Eurojust 1441 υποθέσεις το 2011. Μία μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι που είχαμε 1421 υποθέσεις. Σε σχέση πάντως με πέρυσι, με το 2010 μάλλον, είχαμε περίπου αύξηση των συντονιστικών συνεδριάσεων κατά 45%, σχεδόν διπλασιασμό δηλαδή των συνεδριάσεων. Γιατί τέτοιου είδου συντονιστικές συνεδριάσεις γίνονται μόνο από τη Eurojust. Είναι πολύ σπάνιο να έχουμε στην ίδια τράπεζα ανακριτές, εισαγγελείς από διάφορα κράτη και τους προσκαλούμε να μας δώσουν πληροφορίες για τρέχουσες ε, ανακρίσεις, ε, διώξεις και γίνεται μια ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να καταρτιστεί μια στρατηγική δίωξης. Έχουμε ε, το δίκτυο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών σε πέντε χώρες. Και εκεί ζητούμε ανάμειξη και συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από αυτές τις πέντε χώρες. Έρχονται λοιπόν στη Eurojust, γίνονται συνεδριάσεις με διερμηνία και όπως και η Europol έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου οι πληροφορίες να οδηγήσουν σε συγκέντρωση τεκμηρίων και αποδεικτικών στοιχείων και να, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δικογραφία ουσιαστικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο της Eurojust γιατί όταν έχουμε δίκτυο με πέντε χώρες αποφελούνται όλες από τις γνώσεις που συγκεντρώνονται στη διάρκεια μιας δίωξης. Πρόκειται για πολύ μακρόπνοη προσπάθεια. Και έτσι κάθε χώρα δεν επικεντρώνεται μόνο στην εσωτερική διοκτική διαδικασία, αλλά έχει μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Και έχουμε και στοχευμένη ενίσχυση ε, των δράσεων αυτών Έχουμε ε, συμμετοχή αστυνομικών που κάνουν ε, κατοίκον διερευνήσει, μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών σε αυτέ τι πέντε χώρε του δικτύου για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Και έτσι δίνουμε ένα σαφέ μήνυμα προ του εγκληματίε. Γιατί αυτοί είναι οργανωμένοι, αλλά βλέπουν ότι και εμεί είμαστε εξίσου οργανωμένοι και συντονισμένοι. Και μπορούμε με πολύ αποτελεσματικό τρόπο να αντιδράσουμε και να διώξουμε τέτοιου είδου εγκλήματα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε ως Eurojust και μόνο χάρη στο συντονισμό θα το καταφέρουμε. Χάρη σε πολυμερή δικαστική συνεργασία και συντονισμό. Μπορούμε να έχουμε και διμερή επαφή με φαξ, με κινητά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά αυτό είναι διμερές από μία χώρα σε άλλη. Είναι πολύ περιορισμένο. Ενώ η Eurojust ε, εξασφαλίζει μία πιο ευρεία προσέγγιση, την προσέγγιση Omnibus όπως τη λέμε, και προσκαλούμε όλες τις χώρες ε, ενημερώνονται για το πρόγραμμα έγκαιρος, οπότε έρχονται προετοιμασμένοι και μας δίνουν ε, μια σαφή εικόνα για την ε, ανάκριση τη δίωξη που γίνεται σε μια χώρα και κοινοποιεί τα στοιχεία στους υπόλοιπους. Νομίζω ότι έτσι είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. υπάρχουν διάφοροι τρόποι ε, για να χειριστούμε το θέμα. Όλα είναι δυνατά. Όπως το Ευρωπαϊκό Ένταλμα, για παράδειγμα. Πάντως, κάθε διοκτική διαδικασία χρήζει διαφορετικής προσέγγισης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το συγκεκριμένο εγκληματικό κύκλωμα υπάρχει, για όλα τα εγκληματικά κυκλώματα υπάρχει μία συνταγή για κάθε ξεχωριστή εγκληματική δραστηριότητα υπάρχει ξεχωριστή συνταγή. Πάντω, επαναλαμβάνω, οι συντονιστικέ συνεδριάσει έχουν αυξηθεί κατά 45%, κάτι που είναι πολύ ευχάριστο γιατί δείχνει ότι τα κράτη-μέλη προσφεύγουν στη Eurojust για τέτοιου είδου ε, ε, δικαστικού συντονισμού. Και μάλιστα ε, σε 70% των περιπτώσεων πάνω από τρει χώρε αναμειγνύονται σε αυτές τις διώξεις. Οπότε δεν έχουμε διμερείς μόνο επαφές, μόνο διμερείς υποφέσεις με δύο χώρες, αλλά έχουμε με πολύ περισσότερες τρεις, έξι και χώρες. Και μας ενδιαφέρουν οι δραστηριότητες που γίνονται σε πάνω από πέντε χώρες. Μερικές φορές και εξοκοινωτικές. Κάτι άλλο θετικό είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ε, είχαμε πέρυσι 80% ε, των περιπτώσεων αναφέρονται στους τομείς προτεραιότητας. Γνωρίζετε ποιε είναι οι προτεραιότητε του Συμβουλίου. Ε, σωματεμπορία, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, διαφθορά, απάτη, λεύκαση χρήματο, κυβερνοέγκλημα και τρομοκρατία. Αυτέ είναι οι προτεραιότητε που εντόπισε το Συμβούλιο. Οπότε τα αιτήματα συντονισμού προ τη Eurojust θα φέρουν κυρίω αυτού του τομεί προτεραιότητα. Βέβαια, εξορισμού όλα αυτά τα θέματα έχουν, διασυνοριακά, έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και de facto. Ε, αφορούν περισσότερες από δύο-τρεις χώρες. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει αυξηθεί η ποσότητα των υποθέσεων, αλλά και η ποιότητα βελτιώνεται χάρη στον καλύτερο συντονισμό. Και επίση η ταχύτητα βελτιώνεται, γιατί θα... είναι τόσο σαραγδαίες ε, οι εξελίξεις και τόσο ε, α, ταχύες οι κινήσεις των εγκληματιών που θέλουμε και εμείς αντίστοιχη άμεση αντίδραση και ταχύ αντίδραση των διοκτικών αρχών. Και μάλιστα πέρυσι είχαμε και μια διαδικασία δικαστικής δράσης νέα με ε, κέντρο επιχειρησιακής συνεργασίας, ένα, μια μορφή δικαστικής α, ε, συνεργασίας και συντονισμού. Γιατί έχουμε τέτοιες συντονιστικές συνεδριάσεις, εκεί ε, αποφασίζουμε για μια στοχευμένη ενίσχυση και βοήθεια και στη διάρκεια αυτής της ενίσχυσης, της στοχευμένης, η διεκτικές αρχές των ενδιαφερομένων χωρών συναντιόνται σε 6 ώρα το πρωί σε ένα κέντρο αντιμετώπισης κρίσης. Οπότε με βίντεο διάσκεψη και με μία ενιαία διεύθυνση mail με μία ενιαία τηλεφωνική γραμμή μπορούν να επικοινωνήσουν με τις δεκτικές αρχές των πέντε χωρών. Επίσης έχουν ε, επαφή και με τη Europol και λαμβάνουν τις πληροφορίες από πρώτο χέρι. Μπορούν έτσι καλύτερα να συντονιστούν με αυτό το επιχειρησιακό κέντρο αντιμετώπισης κρίσης, να διασταυρώσουν τις πληροφορίες και να δουν τι χρειάζεται για άμεση αντίδραση. Χρειάζεται ένα νέο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ε, χρειάζεται μια νέα υποβολή αίτησης, αλλά έχουν άμεσες επαφές με τις ενδιαφερόμενες χώρες. Ένα νέο σύστημα εγκαινιάστηκε πρόσφατα και πιστεύω ότι χάρη σε αυτό θα γίνουμε ακόμη πιο αποτελεσματικοί. Εν συντομία θα σας παρουσιάσω δύο υποθέσεις γιατί εμπράκτος μπορούμε να δείξουμε καλύτερα τη λειτουργία μας. Μια σουηδική υπόθεση η οποία ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια και η οποία πραγματικά ολοκληρώθηκε στις 8 Μαρτίου του 2012 όταν ξεκίνησε η δίκη ενώπιον του Σουηδικού Δικαστηρίου. Ξεκίνησε με ένα δίκτυο πολύ οργανωμένο στον τομέα των ε, ναρκωτικών. Ξεκινούσε από την ε, Σουηδία, τη Γαλλία και την Ισπανία με διακλαδώσεις σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κολομβία, Ανδόρα, Βενεζουέλα και άλλες. Ήταν προφανές ότι χρειαζόταν συντονισμός ο συντονισμός ξεκίνησε το 2008-2009, ξεκίνησε η ομάδα έρευνας αφού συστάθηκε 1,4 τόνοι πολύ καλής ποιότητας κοκαίνης και 13 συλλήψεις έλαβαν χώρα, ενώ συνεχίστηκαν ε, μέχρι το Δεκέμβριο του 2010 οι έρευνες. Και τελικά η σύλληψη του επικεφαλής στα σερβικά σύνορα. Ήταν Σουηδός, κάποια μέλη της ομάδας του ζούσαν στην Ελβετία. Υπήρχαν και κάποια παράλια δίκτυα, τα οποία τελικά φάνηκε ότι είχαν και αναλάβει και την νομιμοποίηση των χρημάτων αυτών που προερχόταν από αυτές τις παράνομες διαδικασίες. Ζούσαν σε πολυτελείς βίλες, είχαν σκάφη και βεβαίως όλα αυτά μας ε, βοήθησαν και μας αποκάλυψαν και κάποιες άλλες διακλαδώσεις. 12 εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν σε ακίνητες, επενδύσεις ακίνητης περιουσίας. Έξι από αυτά τα εκατομμύρια κατασχέθηκαν ε, από την περιουσία που δημεύθηκε. Επίσης, 468 εκατομμύρια σε αξία εμπορεύματος επίσης κατασχέθηκε από τις ε, ευρωπαϊκές δυνάμεις. Η Europol, η Europol εργάζεται για μας, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο όσον αφορά την ανάλυση των στοιχείων που βρίσκονται. Μας διευκολύνουν επίσης όσον αφορά την ε, κατάσχεση και την δίμευση περιουσιακών στοιχείων. Αυτό ξεκίνησε, όπως είπα, το 2008, συνεχίστηκε μέχρι το 2012 και εμείς ήμασταν, αν θέλετε, σε επίπεδο δικαστικής συνεργασίας, νομικής αρρωγής, δικαστικής αρρωγής εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλάβαμε επίσης και όσον αφορά την επιλογή των σωστών ε, ε, δικαστικών αρχών, εισαγγελικών αρχών. Γιατί όπως καταλαβαίνετε πρόκειται για πολύ δύσκολους και βαρύς μηχανισμούς και δύσκολο συντονισμό. Καταλαβαίνετε ότι ενεπλάκησαν ε, εκτός της Eurojust και οκτώ κράτη κάτι που μας επέτρεψε να ξεκινήσει η δίκη. Περιμένουμε βεβαίως το αποτέλεσμα της διαδικασίας, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν είχαμε υιοθετήσει την παραδοσιακή οδό τη διμερή Σουηδία-Ισπανία, διμερής επικοινωνία, Σουηδία-Γαλλία, Σουηδία-Κολομβία, η διαδικασία θα είχε πάρει πολύ περισσότερα χρόνια. Γι' αυτό και χρησιμοποίησαμε εμείς την ε, δική μας πολύ πιο γρήγορη και αποτελεσματική συνεργασία. Άλλη υπόθεση, λαθρεμπόριο τσιγάρων από Ουκρανία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ουκρανική, αν θέλετε, καθοδήγηση μέσω της Τσεχίας, Σλοβακίας, Σλοβακίας, Ιταλίας, Γερμανίας Υπήρχαν διάφορες ε, εικονικές εταιρείες με εικονική δραστηριότητα, η οποία ουσιαστικά ακολουθούσε μια εικονική εμπορική συναλλαγή και οδούς. Τελικά όμως ο σκοπός ήταν αυτά τα τσιγάρα να περνούν μέσω από τις, ε, τους συνοριακούς ελέγχους και να φτάνουν στο Ενωμένο Βασίλειο. Υπήρξε λοιπόν εδώ μία συνεργασία ταυτόχρονη έτσι ώστε να μπορέσουμε να χτυπήσουμε και να χτυπήσουμε με καθοριστικό και κέριο πλήγμα τον στόχο μας, τον Ουκρανικό στόχο. 21 Ιουνίου επετεύχθη αυτό. Πώς έγινε αυτό μέσω των νέων κέντρων επιχειρησιακού συντονισμού, κάτι το οποίο όπως σας είπα είναι καινούριο, είναι αποτελεσματικό. Έξι διαφορετικές αρχές συμμετείχαν και χρησιμοποιήθηκαν βεβαίως εδώ και τα μέσα που διαθέταμε από την Europol. Διοκτικές αρχές, δικαστικές, ε, δικαστική συνεργασία ήταν πραγματικά μία πολυμερής, αν θέλετε, συνεργασία για την καταπολέμηση αυτού του δικτύου λαθρεμπορίου τσιγάρων. Την ημέρα την συγκεκριμένη που επιλέγετε για να ξεκινήσει η διαδικασία, καταλαβαίνετε ότι η συνεργασία είναι καθοριστική, η αποτελεσματική, η πραγματική συνεργασία καταρχήν μεταξύ Eurojust και Europol. Και αυτό που είναι πολύ θετικό είναι ότι έχουμε 17 διαφορετικά κέντρα ανάλυσης του Europol που εργάζονται για μας και σε 89 συναντήσεις ε, συντονισμού ήταν παρούσα και η Europol και αυτό είναι κάτι το πολύ θετικό και τώρα πια έχουμε και τη δέσμευση και της Eurojust και της Europol έτσι ώστε να είναι παρόντες σε όλες τις επιχειρησιακές συναντήσεις. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η επιτυχία αυτών των κοινών ε, ε, επιχειρήσεων είναι κάτι που μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις καταπολέμησης της τρομοκρατίας, εδώ καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλες τις δυνάμεις και να έχουμε όλη τη συνεργασία από μέρους των κρατών μελών, αυτό είναι κάτι που πολλές φορές μας περιορίζει. Μπορούμε βεβαίως να έχουμε τα στοιχεία και τα συμπεράσματα της αναλυτικής εργασίας της Europol, δεν μπορούμε όμως να ολοκληρώσουμε την ε, εργασία μας, δεν μπορούμε πολλές φορές να έχουμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση και εικόνα των διαδικασιών μιας τρομοκρατικής οργάνωσης από τη στιγμή που τα κράτη-μέλη περιορίζουν τη δράση μας και επιφυλάσσονται. Κοινέ ερευνητικές ε, ομάδες, κοινέ ομάδες έρευνας υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό και έχουν επιτυχία εδώ και πέντε χρόνια. Γιατί, γιατί εδώ και πέντε χρόνια έχουμε τα τελευταία χρόνια με τη δημιουργία ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων και μετά από την πενταετή πείρα μας με κοινέ συναντήσεις κοινή συνεργασία, οι οποίες οργανώνονται από κοινού και εκ στην Eurojust και στην Europol για την ανταλλαγή συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Αυτές οι κοινέ ε, ερευνητικές ομάδες, κοινέ ομάδες οι οποίες συνεργάζονται, ανταλλάσσουν πληροφορίες, και των οποίων η αποτελεσματικότητα είναι εξαιρετικά σημαντική, όπως είναι σημαντική βεβαίως και η χρηματοδότηση. 2,3 εκατομμύρια είναι η πρικοδότηση αυτών των ομάδων για το 2011. Η Επιτροπή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Επιτροπής έχει εγκρίνει για το παρελθόν αυτήν την δράση. Καταλαβαίνετε όμως ότι αποκλείονται από εδώ και πέρα από τον έλεγχο καθότι δεν έχει ενσωματωθεί κανένας ευρωπαϊκός οργανισμός και ευρωπαϊκή υπηρεσία σε αυτή την πρόβλεψη. Για το 2013 η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι να ζητήσουμε συμπληρωματική χρηματοδότηση και βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι μια συγκεκριμένη επιτυχία. 165 αιτήσει είχαμε πέρσι για τέτοιες κοινέ ομάδες και χρηματοδοτήθηκε η δράση 65 από αυτές στον τομέα κυρίως προτεραιότητας όπως καταπολέμηση λαθρεμπορίου ναρκωτικών και πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολύ συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Θα είναι λοιπόν κρίμα αν δεν συνεχιστεί αυτή η επιτυχής ε, δράση. Μέχρι τώρα βλέπουμε ότι οι διαδικασίες επιταχύνονται και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Εσείς πραγματικά αν μπορείτε και όπου μπορείτε θα πρέπει να στηρίξετε στέλνοντας το μήνυμα ότι θα είναι πολύ κρίμα να μην συνεχίσει αυτή η αποτελεσματική καταπολέμηση του συνοριακού εγκλήματος στην Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον, θα ήθελα να αναφερθώ Στο πολιετές στρατηγικό σχέδιο της Eurojust, ποιες είναι οι μεγάλες κατευθύνσεις, το 2014, η βελτίωση της καταπολέμησης εγκληματικών δραστηριοτήτων και βεβαίως η περαιτέρω εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας. Αν θυμηθείτε τα παραδείγματα που σας ανέφερα μέχρι τώρα, έχουμε διασφαλίσει μια καλή συνεργασία, έναν καλύτερο συντονισμό και περισσότερες δράσεις και πιο αποτελεσματικές δράσεις με τα επιχειρησιακά κέντρα συντονισμού. Τώρα, όσον αφορά τους διάφορους οργανισμούς μας, το κολέγιο της Eurojust και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Επιτροπή σας και την σημαντική νομοθετική εργασία σας. Ναι, να σας υπενθυμίσω, λέει ο Πρόεδρος, μην ξεχάσετε ότι έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο. Εχθές ξεπεράσαμε το μας, Όπως καταλαβαίνετε έχουμε διερμηνία μέχρι τις 12.30. Μην το ξεχάσετε αυτό για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε και κατόπιν να ακολουθήσουν και κάποιες ερωτήσεις από τα μέλη. Ναι, ναι, βεβαίως. Πρόσφατα λοιπόν αντιμετωπίσαμε διάφορες προκλήσεις. Η αναθεωρημένη απόφαση του Συμβουλίου το 2008-2009 θα πρέπει να είχε εφαρμοστεί μέχρι τον Ιούνιο του 2011. Όλα τα κρατημέλη έπρεπε να την υλοποιήσουν, αλλά κρατημέλη δεν την έχουν υλοποιήσει ακόμα. Σε αυτήν την απόφαση του Συμβουλίου υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά άρθρα, το 12 και το 13 το 12 αναφέρεται στο ENCS, δηλαδή συστήματα συντονισμού και το 13 που αναφέρεται στα συστήματα πληροφοριών, ιδιαίτερα βεβαίως υπό κάποιες προϋποθέσεις, όπως παραδείγματος χάνει σε περιπτώσει εμπορίας ανθρώπινων όντων ή σε άλλου είδους παράνομες δραστηριότητες από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας στη Eurojust, πήραμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασίας για τα άρθρα 85, 86, 81 της συνθήκης της Λισαβόνας για τον επιχειρησιακό συντονισμό. Συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των οργανισμών και των υπηρεσιών Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε συνειδητοποιήσει ότι όταν ξεκινήσαμε πριν από 8-9 χρόνια με 80 άτομα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Σήμερα είμαστε βεβαίως περισσότεροι, 300 με το διοικητικό μας συμβούλιο, και βεβαίως η αποτελεσματικότητά μας ε, έχει κάποιους περιορισμούς λόγω και του αριθμού των ε, συνεργατών της Eurojust. Εδώ λοιπόν χρειάζονται διάφορες διευθετήσεις και θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του καλύτερη διαχείριση των θεμάτων και καλύτερη αποτελεσματικότητα, αναδιάρθρωση της διοίκησης και βεβαίως μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου, του Κολεγίου όπως το λέμε και βεβαίως των εθνικών εκπροσώπων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό καθότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των αποφάσεων. Επαναλαμβάνω το άρθρο 85, το άλλο 86 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Από 2009, από το Δεκέμβριο, έχει γίνει πολλή ανάλυση, σκέψη για το τι πρέπει και τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά την ε, αξιολόγηση ε, της δραστηριότητας της Eurojust μέσω των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη διάρθρωσή μας, τη δομή μας, έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Τι αλλαγές διαθωτικές πρέπει να γίνουν για να βελτιώσουμε τη δράση μας. Και βεβαίως συνεχίζουμε από το Δεκέμβριο του 2009 μέχρι σήμερα την ανάλυση των άρθρων 85 και 86. Το άρθρο 86 επίσης το επεξεργαζόμαστε περαιτέρω και Είχα απαντήσει σε μια προφορική ερώτηση της Επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε συναντήσεις με την ε, Εισαγγελική Αρχή όσον αφορά τη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και ποια θα μπορούσε να είναι εδώ η συνεργασία της Eurojust, η εμπλοκή της Eurojust. Εμείς πραγματικά περιμένουμε κάθε είδους ε, πρόταση σύσταση για την αποτελεσματικότερη δράση μας σε όλους τους τομείς, το πάγωμα περισσοιακών στοιχείων, στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης ε, χρημάτων από τις παράνομες διαδικασίες, λεύκανση χρήματος και βεβαίως εσείς σαφώς και με τα εθνικά κοινοβούλια θα παίξετε το ρόλο του αξιολογητή του εκτιμητή της δράσης της Eurojust. Είναι λογικό να ελέγχεται και ο διευθυντής. Το ερώτημα είναι, θέλετε κάτι παραπάνω, θέλετε περισσότερα στοιχεία για να μπορέσετε να είστε σε θέση να αξιολογήσετε τη δράση μας. Ζητήστε, ζητήστε μας αυτά που θέλετε και εξηγήστε μας τι περιμένετε από μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δείξατε πραγματικά αποφασιστικότητα, δέσμευση. Πραγματικά έχετε εργαστεί στη Eurojust και έχετε εργάζεται εκεί από τότε που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια εδώ και 10 χρόνια. Και δείξατε εσείς όλη τη δυνατότητα που έχετε να αναπτύξετε αυτά. Και βλέπω ότι υπάρχει και πάθος, θα έλεγα, για αυτή τη στιγμή, γιατί ε, με πάθος παρουσιάσατε τις απόψεις για το θέμα της ατζέντα τη σημερινής διάταξη. Ούσα πρόεδρος αυτού του σημαντικού σώματος το οποίο συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Νομική Επιτροπή και με τη δική μας Επιτροπή η οποία συνεργείται μετά από την προσπάθησα το, της λησβονοποίησης του τρίτου πυλώνα των κεκτημένων. Europol, Eurojust και περαιτέρω ανάπτυξη δηλαδή σαν το έμβριο θα λέγαμε της υποτιθέμενη ε, σε ένα δημόσιο κατήγορο, δημόσιο εισαγγελέα, ο οποίος θα είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κάνοντας αυτά τα πράγματα να λειτουργήσουν. Αυτό είναι στα σκαριά ακόμη και θα μπορέσει να λειτουργήσει πέρα από τα σύνορα. Νομίζω πραγματικά οι σωστοί άνθρωποι θα έχουν και στη διαδικασία. διαδικασία. Λαμπρά έχουμε τους συνομιλητές, του συμβουλευτέ, που θέλουν να πάρουν το λόγο παρακαλώ. Έχετε το λόγο κύριε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ καταρχήν την κυρία Κόνιξη για την παρουσίασή τη για το πάθο το οποίο επέδειξε στην παρουσίαση, καθώ επίση και για την εκλογή τη στο Eurojust. να ήμουν πολύ επιφυλακτικό πρέπει να ομολογήσω ότι όσον αφορά τα γεωργιαστικέ πραγματικά πώ και κατά πόσο τα χρήματα που κατατίθενται εκεί θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την περίπτωση αυτή. Τώρα είμαι πεπισμένο ότι έκανα λάθο, ότι πραγματικά είναι άξιο ο μισθό αυτών που ασχολούνται εκεί. Εάν δούμε πραγματικούμε τι προτεραιότητε, τα θέματα που θέσατε μέσα στην έκθεσή τώρα, δεν βλέπω καν το, τη, λαθρομεταν... Ε, τη λαθροεμπορία εμπόριο ανθρώπων, λαθεμπορία ανθρώπων. Υπάρχουν, ξέρετε, πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι πνίγονται στις θάλασσες. Sorry. Ε, ότι υπάρχει αυτό το εμπόριο των ανθρώπων, ε, υπάρχει αυτό το λάθρεμπόριο. Ναι, Και τι ακριβώς κάνει το Justice είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί γενικά. Πρέπει, αν το κάνουμε, πρέπει να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί καταλικάζοντας και καταδιώκοντας καλύτερα τους εγκληματίες εκείνου, οι οποίοι ασχολούνται με το εμπόριο των ανθρώπων. Διότι πρόκειται περί ζωών που πρόκειται και ανθρώπων που χάνονται στη θάλασσα. Σε ένα άλλο σημείο φτάσατε να πείτε ποιος θέλει να αλλάξει αυτά τα πράγματα πρέπει και τελειώστε ε, με μια θετική νότα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ε, είμαστε πάντοτε ανοιχτοί και για αυτά τα οποία έχετε στις πρωτεΐνες και σας ευχόμεθα καλή επιτυχία. Κυρία Ζίκελ παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να συγχαρώ για, τις νέες, για τα νέα σας καθήκοντα και λυπάμαι ότι είμαστε ευάρυθμοι σήμερα. Το Eurojust, Eurojust είναι ένα θεσμικό όργανο πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με τη συνεργασία στο ποινικό επίπεδο και στην έκθεσή σας μας είπατε πάρα πολύ σαφώς για την εξαιρετική σημασία που έχει η συνεργασία αλλά και ο συντονισμός υποθέτει ότι όλοι μετέχοντας θα δείχνουν την καλή διάθεση και ότι όλοι θέλουν να φτάσουν ομού σε μια, σε μια επιτυχία έκταση για να είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή, καλό αυτό το αποτέλεσμα, το κοινό αποτέλεσμα. Θα ήθελα λοιπόν να ασπαστώ την αισιοδεξία με την οποία εσείς παρουσιάσατε τα πράγματα, αλλά δεν είμαι καθόλου πεπισμένη ότι πραγματικά οι αρχές, οι αστυνομικά όργανα, οι αστυνόμοι αυτοί καθ' ασπάζονται αυτή, αυτό τον, την αισιοδοξία. Κατά πόσο πραγματικά είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν ορισμένε αρμοδιότητες που έχουν για να εργαστούν μαζί, για να συνεργαστούν, για να έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ο όπως Βουζουτή μα είπε προηγουμένω ήταν λίγο λιγότερο αισιόδοξο και θετικό από αυτό που σκεφτόταν, που, ε, που είχε κατά νου καλύτερα και ότι τα πράγματα, το επίπεδο της εφαρμογής ήταν πάρα πολύ περιορισμένο. Έρχομαι όμως στο θέμα του συντονισμού. Ο συντονισμός για τη μεγάλη εγκληματικότητα, ε, ναρκωτικά, ε, δουλεμπόριο. Πιστεύετε ότι οι πρωτοβουλίε τέτοιου είδους μπορούν να ληφθούν και ότι αυτές είναι απαραίτητες και κατεπήγον χαρακτήρα για να υποχρεώσουμε τα κάτι μελη να συνεργαστούν. Μία τέτοια πρωτοβουλία εκ μέρου του Eurojust θα ήταν υπεραπαραίτητη για να υπάρχει πραγματικά ένα δικαστήριο, να υπάρχει ένα εισαγγελέα. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα μπορούσε ενδεχομένω να έχει μια διάσταση πιο ευρωπαϊκή για την καταπολέμηση, για την καταπολέμηση της μεγάλης και μια τελευταία ερώτηση όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα. Το θέμα αυτό, όπως ξέρετε, δεν ε, την χάνει ευρέας στήριξη ε, εδώ στο Κοινοβούλιο και θα ήθελα να μου πείτε πώς αντιμετωπίζει αυτό στην Eurojust. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα στην πράξη ρεαλιστικά, γιατί ξέρω ότι τα διάφορα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν εντελώς διαφορετικά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. κυρία Ματιό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλά θορίσατε κυρία μου, κυρία Πρόεδρε και συγχαρητήρια για τα αποτελέσματα τα οποία έχετε λάβει. Δεν, ασπάζουμε την απόψη των συναδέλφων και Eurogist και οι αρμοδιότητες οι οποίες ανέλαβε και οι οποίες είναι ενισχύει εδώ και πέντε χρόνια μόνο δεν νομίζω ότι αξίζει να διορθωθούν πιστεύω τα αποτελέσματα τα οποία έχει μέχρι στιγμή θα επιτρέψει στα κρατη μέρη γιατί όλα δεν συμμετέχουν θα τα επιτρέψει λέω να το κάνουν και να υπάρξει μια συνεργασία. Ο Σάιμον το είπε προηγουμένω ότι υπάρχουν ορισμένοι τομεί οι οποίοι δεν είναι ανοιχτοί ακόμη και είναι πιο δύσκολο ενδεχομένω, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διασυνοριακή κλιματικότητα. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί κάποια στιγμή, τόσο λοιπόν στο δικαϊκό όσο και στο αστυνομικό επίπεδο υπάρχει ένα μυστικό το οποίο πραγματικά πρέπει να αρθεί. Είναι δύσκολο βεβαίως, αλλά πρέπει και μπορεί να γίνει. Καλό κουράγιο να έχετε λοιπόν κυρία Πρόεδρε, διότι θα χρειαστεί χρόνος για να το κατορθώσουμε αυτό. Τι σκέπτεστε και τι φρονείτε όσον αφορά τον Ευρωπαίο εισαγγελέα. Νομίζω θα δυσκολευτούμε για να αυτό για να γίνει δραστήριος και αποτελεσματικός και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον κατορθώντε εσείς έχετε πληροφορίες για τα σωστά αποτελέσματα τα οποία δημιουργούνται. Παραφερθήκα σε ένα παράδειγμα. Κατά πόσο πραγματικά γυρνάτε στα διάφορα κράτη-μέλη για να δείτε ε, πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα, πώς γίνεται αυτή η συνεργασία και αυτός ο συντονισμός, επιτόπου δηλαδή. Και όσον αφορά την τρομοκρατία, μας είπατε προηγουμένω ότι έχετε κάποια δυσκολία να έχετε ε, συνεργασία με την Europol κατά πόσον είναι αποκλειστικότητά του, είναι κλειστά εντό εισαγωγικών τα σύνορα με αυτού, οι σχέσει σα. Ευχαριστώ κύριε Βακεντάη, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την κυρία Κόνιγκς για την παρουσίαση που μας έκανε. Να συγχαρώ και εγώ ε, την κυρία Κόνιγκς για το διορισμό της, όπως και οι συνάδελφοι. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Και εγώ είμαι υπέρ της ιδέας του συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητο ο συντονισμό για την πάταξη σοβαρών και διασυνοριακών εγκλημάτων. Η ομάδα μου είναι κατά της ιδέας για μια ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή. Η συνεργασία και ο συντονισμός κατά τη γνώμη μας δεν σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκχωρήσουν τα τις εξουσίες τους. Ίσα ίσα με την ισοτιμισμό και τη συνεργασία ενισχύονται οι δραστηριότητές τους. Έχω δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρόσφατα παρευρέθηκα σε μια διακοινοβουλευτική συνεδρίαση στην πατρίδα μου με μέλη της Βουλής των Λόρδων, της Βουλής των Κοινοτήτων και ευρωβουλευτές. Και ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα. Μιλήσατε εσείς για την για το συντονισμό και συνεργασία Europol και Eurojust, εμείς ασχοληθήκαμε με τη Europol. Κάποιος από τη Βολή των Λόρδων είπε ότι χρήσιμο θα ήταν να συμπίπτει η δημοσίευση των εκθέσεων της Eurojust με την Europol για να μπορέσουμε να εξετάσουμε από κοινού τις δραστηριότητες και των δύο οργάνων. Μπορείτε να το λάβετε αυτό υπόψη. Μία άλλη ερώτηση. Στο παρελθόν πρωτοστατήσετε σε διώξει κατά τρομοκρατών και οργανωμένων κλίματος. Ποια είναι λοιπόν η γνώμη σα ω επαγγελματία για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διακοπή των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία PNR του Μητρώου Ονομάτων Επιβατών. Ευχαριστώ. Κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ. Δεν είμαι και ο πιο ε, ένθερμος ζηλωτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε καν της Eurojust. Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να έρχομαι στις συνεδριάσεις και να ε, εξετάζω τα πράγματα αντικειμενικά. Αναφέρεται προηγουμένως στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ επιβαχό το ζήτημα αυτού του ενδάλματος, γιατί έχασαν ε, τις εξουσίες τους, τις δικαιοδοσίες τους σε δικαστήρια και κυρίως στο ανώτατο δικαστήριο που δεν μπορούν να ε, προβούν σε έκδοση για λόγους ε, ανεπαρκούς ε, τεκμηρίωσης. Βέβαια, εσείς είναι ένα εργαλείο που διαλέγετε, δεν, το ένταλμα δεν είναι δική σας αρμοδιότητα η έκδοσή του. Θεωρείτε ότι η Eurojust αυτές τι ε, τις συντονιστικές συνεδριάσεις εξετάζει με επικριτικό τρόπο τα τεκμήρια που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη πριν εκδοθεί ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη ανεξάρτητα από τη χώρα που θα το εκδώσει. Με άλλα λόγια, γίνεται δεύτερη εξέταση των ε, ε, αποδεικτικών στοιχείων ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια των ε, εξουσιών ε, που παρατηρήσαμε όταν ε, αποφασίστηκε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Βλέπετε τελικά δεν είμαι και πολυ απεσιοδοξος απεσιόδοξο, είμαι μάλλον αισιόδοξο. Κυρία Κόνιγκς, 5-10 λεπτά σας έχουν απομείνει. Σας θέλω, παρακαλώ να ολοκληρώσετε εγκαίρως για να μην έχουμε πάλι υπέρβαση του ωραρίου όπως χθες κάνετε κάποιες γενικές παρατηρήσεις αν μπορείτε και αναφερθείτε στο πιο ενδιαφέρον σημείο που είναι ο συντονισμός της Eurojust με τη Europol. Γιατί και η Europol ασχολείται με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και ελπίζουμε να βελτιωθεί η λειτουργία της στο μέλλον με την κοινή δικτύωση και την καλύτερη ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των δύο οργανισμών, της Eurojust και της Europol. Επίσης, ε, υπευλήθη ένα σχόλιο για την ε, δυνατότητα βελτίωσης της επικοινωνίας. Το έχουμε δει πολλές φορές. Όλες οι βελτιώσεις που έγιναν στον ΕΟΧ δεν φτάνουν στα αυτιά των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν υπάρχει προβολή τους υπάρχει ένα επικοινωνιακό κενό. Γιατί κάνουμε ό,τι μπορούμε και έχουμε σημαντικά επιτεύγματα σε ό,τι αφορά την ε, εξυπηρέτηση των πολιτών και την πάταξη του διασυνοριακού εγκλήματος, αλλά δυστυχώς οι πολίτες το αγνοούν, γιατί δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Ακόμη και οι εισαγγελείς ή δικαστές των χωρών μελών δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες που έχουν και το τεράστιο δυναμικό που υπάρχει για συντονισμό και συνεργασία. Δεν ε, γνωρίζουν καν τις προοπτικές ε, περαιτέρω εξέλιξη αυτών των σημαντικών εργαλείων. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ενημερωθούν καλύτερα οι εισαγγελείς, οι διοκτικές αρχές, οι δικαστές, αλλά και ο κόσμος για τις δυνατότητες που υπάρχουν. Ευχαριστώ. Πόσα δευτερόλεπτα μου έχουν μείνει για να απαντήσω όλες αυτές τις ερωτήσεις το συγγνώμη από τους διερμηνείς άμα κρηγορήσω. Θα κάνω ό,τι μπορώ πάντως να ολοκληρώσω σύντομα. Κύριε Μπουσουτήλ, φυσικά πρέπει να επιτελέσουμε σωστά το έργο μας και να πείσουμε γι' αυτό και εξαρτώμαστε από τα αιτήματα των κρατών μελών. Αν τα κρατημέλη δεν έχουν πιστεί για την αξία της Eurojust, δεν θα απευθύνονται σε αυτήν. Και έχουμε και κάποιες ευθύνε. Ε, γιατί όντως κάνουμε πολλά, πολλή δουλειά, πολύ επικοδομητικό έργο, αλλά δεν το διαφημίζουμε παρκώς. Ε, επικοινωνιακά κάπου χωλένουμε. Αυτό είναι δική μας ευθύνη. Να προβάλλουμε περισσότερο το έργο μας, που όντως είναι πολύ σημαντικό. Πάντως, Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η επικοινωνία επιδέχεται βελτίωση. Όντω, η προβολή θα πρέπει να βελτιωθεί. Η προβολή του έργου τη Eurojust. Δεν γίνεται αρκετή διαφήμιση. 50% του έργου μα παραμένει άγνωστο, στην αφάνεια. Βέβαια, είναι λογικό γιατί έχουμε να κάνουμε συνεργασία δικαστικών αρχών, οπότε υπάρχει και το, η εμπιστευτικότητα, το απόρριτο μερικών πληροφοριών, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να προβάλλουμε κάποια έργο μα. Μερικές φορές χρειάζεται να περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα και εκεί είναι η σημαντική ισορροπία που θα πρέπει να βρούμε. Πάντω, χαίρομαι για την αισιόδοξη σα τελική παρατήρηση. Ούτε κι εγώ θέλω να είμαι απεσιόδοξη, ούτε αρνητική. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω τυφλό και ότι αγνοώ τα προβλήματα. Όντω ένα πρόβλημα που έχουμε είναι στην επικοινωνία. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την επικοινωνιακή μας στρατηγική προς τους ενδιαφερόμενους. Και οι βασικοί ενδιαφερόμενοι είναι τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει προς αυτά να βελτιώσουμε την επικοινωνιακή μας πολιτική. Το θέμα της εμπορίας των ανθρώπων εμπίπτει στο THB, στις βασικές προτεραιότητες. Εμπίπτει λοιπόν και η εμπορία των ανθρώπων σε αυτό που είπατε γιατί είχαμε ένα παράδειγμα εμπορίας, σωματεμπορίας στην Γαλλία, στην οποία συνδέονταν 10 ε, χώρες και περνούσαν από τα νησιά της Μάχης. Μερικές φορές ε, άνθρωποι πληρώνουν τεράστια κονδύλια για να μεταφερθούν και μάλιστα σε τελείως απάνθρωπες και ξεφτυλιστικές συνθήκες. Και είχαμε ε, επαφές με της κεντρικές αρχές της Γαλλίας αλλά και με άλλες χώρες προκειμένου να βελτιωθεί η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Αλλά εμείς εξαρτώμαστε από τα κράτη-μέλη. Δεν αποτανθούν σε εμά, δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη αυτό το πρόβλημα. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση της κυρίας Σίπελ, Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για την επίσκεψη σας τον Οκτώβριο. Βεβαίως χρειαζόμαστε διάλογο, χρειαζόμαστε δεσμεύσεις, αμοιβαία κατανόηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε και το περιμένουμε. Είναι καθοριστική η ενημέρωση. Δεν μπορεί κανείς να ξεκινήσει συντονισμό αν δεν έχει βασικές πληροφορίες. Και αν κάποιος πάει στο άρθρο 85 της συνδέξη Λισαβόνας. Δεν αναφέρομαι τώρα στο πραγματικό κείμενο, ερμηνεύω. Πρόκειται για την καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος βάσει πληροφοριών που δίνονται από τα κράτη-μέλη και από τη Europol. Είναι εξίσου σημαντικές οι δύο πηγές, τα κράτη-μέλη και η Europol. Αν δεν ενισχύσουμε λοιπόν την συλλογή πληροφοριών από μέρους της Eurojust, θα περιμένουμε μονίμως την παράκληση των κρατών μελών. Και εδώ αναφέρομαι στην απόφαση που θα υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να στείλουν πληροφορίες και στη Eurojust και στη Europol. Είμαι αρμόδια για την τρομοκρατία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως αυτό οδηγεί σε μια ενίσχυση της παροχής πληροφοριών και αυτή είναι η κατάσταση και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση των διαδικασιών που αφορούν τους τρομοκράτες, σε όποια φάση και αν βρίσκονται αυτές οι διαδικασίες. Και αυτό για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν την τρομοκρατία βάσει της, του άρθρου 13, εάν το άρθρο 13 και το σύστημα συντονισμού σε εθνικό επίπεδο μεταξύ της Eurojust και της Europal, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η πληροφόρηση περνάει, ότι το σύστημα λειτουργεί και τότε θα μπορέσουμε και εμείς να πάρουμε πρωτοβουλίες για συντονισμό και αυτό θα μας βελτιώσει σαφώς τα αποτελέσματα. Δεν θα χάνουμε δηλαδή κάποιες ευκαιρίες γιατί ένα κράτος μέλος δεν απευθύνεται σε εμά. Εγκαίρος. Εμείς δεν μπορούμε, αν θέλετε, να χτυπήσουμε την πόρτα ενός κράτους μέλους για να ξεκινήσουμε μια ε, μακροπρόθεσμη συνεργασία. Επαναλαμβάνω το άρθρο 26. Χρειάζεται ομοφωνία Ομοφωνία όμως δεν θα επιτευχθεί ποτέ, ας είμαστε ρεαλιστές. Γι' αυτό και θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ εννέα κρατών μελών σε κάποιες ειδικέ, αν θέλετε, θεματικές ενότητες και συντονισμός όπου ο ρόλος της ε, Eurojust θα είναι καθοριστικός, είναι ένας ρόλος κλειδί. Η καταπολέμηση αυτών που ονομάζουμε, αν θέλετε, συναφή εγκλήματα. Ναι, νομίζω ότι με κοιτάτε γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, έτσι. Τι να κάνω. Έχετε ένα λεπτό. Δεν θα με λιντσάρουν οι διερμηνείς. Να συνεχίσω. Ε, εμείς λέμε αυτή τη στιγμή ότι θα πηγαίνουμε βήμα προς βήμα όσον αφορά το, βήμα προς αφορά το συντονισμό και νομίζω θα έχουμε αποτελέσματα μέσα αυτό, μέσα από ένα κείμενο και αυτή είναι ο τρόπος με τον οποίο σε αυτό τον ειδικό τομέα, εάν πραγματικά φέρουμε κόσμο ο οποίος τίθεται υποκρίση, αυτός είναι ο τρόπος που θα ακολουθήσουμε. Και νομίζω πως πραγματικά η παρακολούθηση εκ του σε αυτό το θέμα θα πρέπει να μας δείξει πώς επίδε, επί, πώς επιβάλλουμε αυτά τα πράγματα, πώς θα υπάρχουν οι καταδίκες και νομίζω πως επιβαλλουμε αυτα τα πραγματα πως θα υπαρχουν οι καταδικες και νομιζω πως πραγματικα θα μας οδηγήσει σε αυτό το μονοπάτι ακόμη πιο μακριά. Η W ήταν ένα από τα ερωτήματα Υπάρχουν βέβαια πολλά παραδείγματα τα οποία μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή. 16-17 σε περίπτωση που υπάρχει σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο τέτοιων υπάρχει μπορούμε να εκδώσουμε αποφάσεις οι οποίες θα, στοχεύουν προς την αυτή κατεύθυνση καθώς επίσης όταν υπάρχουν όταν δεν έχουν γίνει σεβαστά τα όρια Ψάχνουμε λοιπόν να υπάρξει ταυτόχρονη εκτέλεση αυτών. Στο Μιλάνο ή αλλού σε Σε πέντε μέρες λοιπόν να υπάρξει ένα συντονισμός σε 20 στόχους, οποίους έχουμε κάνει Ρουμανία, Γαλλία, Ιταλία κλπ. Λόγω της αυτού του εντάγματος σύλληψης το οποίο έχει εκδοθεί και Μερικές φορέ βεβαίω. υπάρχει το θέμα ότι δεν, οι διατυπώσει δεν ήταν σωστέ, η γλώσσα δεν ήταν σωστή και υπάρχει έλεγχος ο οποίο γίνεται για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ την κυρία Ματιό για την ερώτηση την οποία μου έθεσε. Αληθεύει πως για τις μικτές για τις επιτροπές ανάκρισης κοινέ ομάδε έρευνα οι οποίε υπάρχουν και πραγματικά υπάρχουν τα χρήματα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτέ και βεβαίω δίνονται δυνατότητα για διερμηνία, ξενοδοχείο και όλα τα θέματα τα οποία αποδομούν αυτό. Εάν πραγματικά περάσουμε σε όλες τις περιπτώσεις και έχουμε όλε αυτέ τι εγκαταστάσει και τι διευκολύνσει, βεβαίω αυτό θα κοστίσει πάρα πολλά Εκείνο που θέλουμε είναι αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια γραμματεία η οποία γραμματεία θα μπορεί στο Eurojust να υπάρχει εγχειρίδιο, υπάρχει ένα Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διάφορες καταρτήσεις, προσπαθούμε να επιδείξουμε κάνοντας το το καλύτερο μπορούμε αυτό και κατά πόσο μπορούμε και εφόσον δεν έχουμε τον Εδώ μπορεί να τελειώσουμε. Νομίζω πως πραγματικά απάντησα για να σας πω. Σας ευχαριστούμε την κυρία Κόνιξ, ευχαριστώ που ήρθε εδώ μια εκθέση η οποία παρουσιάστηκε ενώπιον και ευχαριστώ και σα όλου που ήσασταν εδώ, το Σα ευχόμαστε επιτυχία, δείξατε ότι είστε αποφασισμένοι, δείξατε ότι είστε πεπισμένοι και νομίζω ότι αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το φθινόπωρο θα υπάρχει μια αντιπροσωπεία που θα πάει στη και να σα επισκεφτεί να δείτε με επιτόπου πώ εργάζεστε και κατά αυτόν τον τρόπο να περάσουμε στη λεπτομερή παρουσίαση των πραγμάτων, γνώση των πραγμάτων καλύτερα και σας ευχαριστώ λοιπόν και σας ευχαριστώ όλους. Ε, παραλαμβάνω στις δυόμιση η συνεδρίαση και όχι στις τρεις, στις δυόμιση συνεδρίαση.